Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ανακοινώνω την έναρξη τη ε, συνεδρίαση. Υπάρχουν παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ο Πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει ε, και αν έχετε να κάνετε παρατηρήσει. Περνάμε στα πρακτικά. 7 Δεκεμβρίου του 2015. Έχει διαβάσει κανείς τα πρακτικά. Αν τα έχει διαβάσει κανείς να εκφράσει αντιρρήσεις. Όχι, δεν υπάρχουν εγκρίνσεις. Εγκρίνονται λοιπόν. Και περνάμε τώρα στο 4 της μέσης διάταξης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο συνάδελφος Χάουιτ είναι ο εισηγητής. Μα ποιος τον ε, αντιπροσωπεύει τότε. Ποιος τον εκπροσωπεί. Μάλιστα. Ο συνάδελφος Φλέκενστάιν. Τι πάθαμε.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 Έλεγχος. γιατί την συμβιβαστική 7, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. 29 ψήφοι υπέρ, 3 ε, κατά, 17 αποχές, έγκρινεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές, έγκρινεται. Η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 47 υπέρ, 4 κατά, 0 αποχές εγκρίνεται. Κύριε Φλέκενστάιτ, να πείτε χαιρετίσματα στον εισηγητή. Τέλειο ήταν αυτό. Μόνο συμβιβαστικέ προτάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σα, αλλά είναι πραγματικά φανταστικό. Αυτό καταδεικνύει η ιδανική συνεργασία μεταξύ των σκιωδών και του εισηγητή. Σα ευχαριστούμε λοιπόν. Και περνάμε τώρα στο σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη σε, σε ό,τι αφορά την διακίνηση των ανθρώπινων όντων στι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Λόχμπίλερ είναι η εισηγητρία. Έχετε να κάνετε καμία παρατηρήση κυρία Λόχμπίλερ. Ωραία. Α ψηφίσουμε λοιπόν κατευθείαν στην παράγραφο 1 υπέρ. Συγγνώμη. Τροπολογία 57 στην παράγραφο 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58. Δεν θεωρήθηκε παραδεκτή η τροπολογία αυτή. Δεν ξέρω γιατί. Βάσει του άρθρου 54 θεωρήθηκε μη παραδεκτή αυτή η τροπολογία. ε, δεν είναι μέσα στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Εντάξει, οπότε δεν πρόκειται να ψηφιστεί. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 και 61 που ταυτίζονται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρασε. 28 με 25 απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά απόχε εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Όχι, όχι, είναι σε δύο τμήματα, συγγνώμη. Σε τρία τμήματα μάλιστα. Τμήμα 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής. Πέρας. 28-23 γίνεται δεκτή με τρεις αποχές. Στη συνέχεια, στην τροπολογία 98, λέει ο πρόεδρος. 97 αλλά έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 98. Υπέρ κατά έλεγχος. Πέρας. Απερίφθη. 25-29. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 10 υπέρ κατά αποχές φρέσκο. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 132 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 140 υπέρ. 139 θέλετε έλεγχο. Εντάξει. Ξεκινάμε. Πέρας ψηφοφορίας. 39-14 εγκρίνεται, σαφώς. Ποιος το ήθελε αυτό τον έλεγχο. Εντάξει. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. 141 έλεγχος. Μάλιστα. 19 με 36 απορρίπτεται. Ήταν 141. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 142. Πέρας. Ψηφοφορίες. 27-21. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά απόχε εγκρίνεται, συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, τροπολογία 155 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 156 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 158 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 162. Υπάρχει κάποιο σφάλμα εδώ. 165 λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές. Πάλι. 165 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. 25-30 απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας ψηφοφοριάζει 25 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. 173. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170, 180. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183. Είναι και συμβαστική 18. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχετε κάποιο πρόβλημα κύριε Πέτακλε. Την άλλη φορά να πρέπει να δικαιολογείτε. Είναι το άρθρο 54. Μα τι είναι το 54 λέει ο πρόεδρος. Αυτό όμω μπορεί να το αποφασίζει το προσωπικό, μπορεί να το αποφασίζουν οι υπάλληλοι, κατά πόσο είναι παραδεκτοί ή μη. Ε, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε εμεί. Θα πρέπει οι βουλευτέ να το γνωρίζουν. Συζητήθηκε με τους σκιωτής. Α, μάλιστα. Θα έπρεπε να το έχω διευκρινίσει εξ αρχή. Ναι. Για την έκθεση αυτή υπήρχε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχαμε ε, κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή ΦΑΜ. Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολη η όλη διαδικασία και κάποιες τροπολογίες ε, ψηφίστηκαν, κάποιες άλλες ενσωματώθηκαν στο κείμενο. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους υπαλλήλου των διαφόρων επιτροπών. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως έτσι την πολιτική. Εμπιστεύομαι φυσικά τους υπαλλήλου, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγχονται. Κύριε Λοκμπίλερ. Κοιτάξτε, εμπιστεύομαι τον κύριο Μπούζεκ και αποφασίσαν σε αυτή τη διάσκεψη των Προέδρων να ε, συνεργαστούν σε αυτή τη σύνθεση. Μάλιστα, καλή ιδέα αυτό, αλλά για την άλλη φορά θα ήθελα να πω ότι ο Πρόεδρος και οι συντονιστές θα πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους και τα αίτια. Μπορεί να στέκουν, μπορεί και να μην στέκουν. Ε, θα έπρεπε να είναι ο κόσμος ο οποίος έχει στείλει τροπολογίες θα πρέπει να ενημερώνεται και δεν ενημερώθηκαν. Δεν βλέπετε εδώ, ο κύριος δεν ξέρει. Δεν υπήρξε ενημέρωση ή υπήρξε ενημέρωση με τρόπο μη αποδεκτό. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Ναι. Λοιπόν, τώρα συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Uh, 190. 190 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. βαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 ε, υπέρ, κατά Ξανά. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Για τη 206. επτά. Υπέρ. Κατά. Α, ναι, πρέπει να κλείσουμε την ψηφοφορία για την 206. 21 υπέρ, 35 κατά απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ. Σε χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες έλεγχος, αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας, 25 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 συμβιβαστική. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι η ίδια 29 του τζιπ. Η 30. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 20, συμβαστική 22 υπέρ, κατά Αποχές. Έγκρινεται. Και τώρα περνάμε στην 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά Ξανά για τα 43 παρακαλώ να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. 21 υπέρ, 3 κατά, απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Η 50 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται και αυτή. 51 υπέρ. Κατά. Η 51 λέω υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι πέταλε τροπολογίες δεν είναι παραδεκτές. Οι 96. 56 λέω υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά παρακαλώ την 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας, 28 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Η 1, τροπολογία 1, πέτερλε, υπέρ. κατά αποχές. Στις συντηρητικές σκέψεις θα τον ε, επαναρθώσουμε. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το τρία. για την τρία. Τέλος πάντων. Δείξτε λίγη ευγένεια, συνάδελφοι. Πέρας 33 υπέρ 21 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Πέτερλε, εγκρίθηκε. Οι 2 και 7 καταπίπτουν και άρα πάμε στην 4-8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να συστήσουμε στους Πολωνούς ε, συναδέλφους ε, του ΕΛΚ να ε, ξεχωριστά τις τροπολογίες τους. εγκρίθηκε. 6, 16, 18 και 19. Ταυτόσιμες όλες τους. Να ξέρα ποιος ήταν και ο υπεύθυνος για αυτές. Μάλιστα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Εγκρίθηκαν. Η 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, τώρα το θυμηθήκα. Ε, αυτόματα εγκρίνονται υπό το άρθρο 54 του κανονισμού. Τώρα κατάλαβα τι μου λέγατε. Ε, μα το μόνο που είπα είναι ότι το κατάλαβα. Ότι αυτόματα θεωρούνται εγκεκριμένε. Αλλά δεν βελτιώνει φυσικά την κατάσταση αυτή. Τι είναι το FV. Παράγραφος 3 της Επιτροπής ε, Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Χωρίς... Έχω ε, στην ψηφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Α, είναι πάλι αυτόματη η έκθεση βάσει του άρθρου 54, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Πέτρελε, μην θέτετε τις τροπολογίες σας μέσω της Επιτροπής Γυναικών. Αυτό θέλω να σας συνιστήσω. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγγελό. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Επιτροπής Γυναικών. Ψήφι υπέρ. Παράγραφος 5 καλύτερα. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω ότι Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. 33-21 εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Επιτροπή γυναικών σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 10 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 13 σε τμήματα, σε δύο πρώτο τμήμα κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα πέρας της φοφορίας Η 22-25 απορρίπτεται. Παράδοση 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της ε, παραγράφου 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα της 16 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Η 10 εγκρίνεται. Γνωμοδότηση <clears throat> της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, παράγραφος 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέρας προφορίας ελέγχου. 26-23 εγκρίνεται πράγματι. Παράγραφος, 20, 7 υπέρ. 7 υπέρ. Παράγραφος 7 υπέρ. Κατά. Τι γίνεται τώρα με την παραγωγή 8. Καλύπτεται από τις τροπολογίες του 27 Ντρουά και άρθρο 22 ή όχι. Ψηφίζουμε και θα ελέγξουμε αν έχει καλυφθεί υπέρ της 8 της Λίμπε, παραγωγή 8, κατά έλεγχος. Πέρας προφορίας 45-10. Εγκρίνεται. 10 της ΛΥΜΠΕ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος. Παράγραφος 13 ΛΥΜΠΕ σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 λίμπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίπε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλύπτεται μέρη από τη συμβαστική 20 για την παράγραφο 19, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να ψηφίσουμε το τμήμα το οποίο είναι ακάλυπτο. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς ψηφίζουμε εδώ πέρα. Μπορούμε να ψηφίσουμε όμως παρακαλώ. Να μας εξηγήσετε κυρία εισηγήτρια. Τι δεν καλύπτεται. Ποιο είναι το τμήμα το οποίο δεν καλύπτεται. Λέτε ότι καλύπτεται εν μέρη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι καλύπτεται και τι όχι από τη Συμβαστική 20. Κακή προετοιμασία, λέει ο πρόεδρος. Δεν νομίζω, λέει η κυρία Λόχπιλντερ. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό και να σας διαβάσω το κείμενο, αλλά... Εγώ προτείνω το αφήσουμε εκτός. Πείτε το καθαρά στην Ολομέλεια να φέρουν αυτό το κομμάτι το οποίο δεν καλύπτεται. Αυτό το κομμάτι που δεν καλύπτεται να υποβληθεί ως τροπολογία στην Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στην ΛΥΜΠΕ 20 που καλύπτεται από τη Συμβεστική 12. Αλλά να την ψηφίσουμε. Όχι, καλύπτεται. Και η επόμενη. Λίμπε 21 καλύπτεται. Από την ΦΕΜ 15. Οπότε λίμπη 22, συγγνώμη, λέει κύριε Λόχ Μπίλερ, είναι θέμα διαδικαστικό. Δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο. Λέει ότι είναι μία ένδειξη ότι, ότι υπάρχει ήδη στη συμβιβαστική. Πρόεδρος, αν είναι ήδη μέσα στη συμβιβαστική, η συμβιβαστική είναι ξεχωριστή. Αυτό είναι ε, κάτι που κάνουμε διαρκώς. Οτιδήποτε δεν είναι ε, ξεχωριστό θα πρέπει να υποβληθεί ως τροπολογία στην Ολομέλεια. Ναι, αλλά κάτι καλύπτεται, ένα κομμάτι καλύπτεται στη συμβιβαστική της, ε, στην ΤΡΟΑ και το άλλο στη ΛΥΜΠΕ και τα ψηφίσαμε ξεχωριστά. Να το κλείσουμε, ε, έφερε κάποιος. Yeah, Καλύπτεται συνεπώς. Δεν θέλω να... Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για πράγματα που καλύπτονται ήδη. Πρέπει να καταρτήσουμε άλλο κατάλογο τότε. Εγώ ψηφίζω τη ΛΥΜΠΕ 22 τώρα. Ψηφίζουμε τη ΛΥΜΠΕ 22 τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπ 23 το ίδιο ΛΥΜΠΕ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 ψηφίζουμε το τμήμα αυτό το οποίο δεν καλύπτεται και το οποίο θα εισαχθεί με τη συμφωνία της εισηγητρίας. Ποιος είναι υπέρ του τμήματος που δεν καλύπτεται κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Λίμπη 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπη 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 32 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 33 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 34 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Λίμπε 35. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην NV3. Υπέρ. Κατά. Ξανά, NV3 λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Την 5. NV5 παρακαλώ ελέγχουμε ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Με οριακή διαφορά, πέρα από το κατά. Αστείευεται ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ. Λίγο πιο πολύ... Ναι, έκανα Ενδυνέα, υπέρ. Κατά. Ενδυνέα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένμι 12. Ένμι 10. Το σημείο που δεν καλύπτεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβι 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόεδρε, λέει η συγγητρία, εδώ θα πρέπει να κάνω προφορική τροπολογία. Έχετε καθυστερήσει, σα παρακαλώ. Όχι, έχετε αρχίσει, σα παρακαλώ να είστε προετοιμασμένοι γέρο. Ήταν στον κατάλογο και είχε ανακοινωθεί, όχι στο δικό μου κατάλογο, λέει ο πρόεδρο. Είναι στο δικό μα κατάλογο, να το βάλετε στην ολομέλεια. Είναι τεχνική λεπτομέρεια και θα βελτιούσε. Όχι, δεν το επιτρέπω. Έχετε, το έχετε λάβει ω προφορική τροπολογία, το έχει λάβει κανεί. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες το έχουν λάβει. Κάποιοι όμως εδώ πέρα στην αίθουσα δεν το έχουν λάβει. Έχετε λάβει την τροπολογία αυτή, την έχετε όλοι σας. Μάλιστα, θα την ψηφίσουμε τότε. NB12. Με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Παρακαλώ. Πέρας. 26 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται ως εκ τούτου. NV16 υπέρ. Μη κατά. Άποχες. Δεν συμμετείχε το ΕΛΚ, άρα εγκρίνεται. Δεν ψηφίσατε, δεν συμμετείχατε. 21. Τροπολογία 21. Υπέρ. nv 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. έγκρινεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. έγκρινεται. 24. Το τμήμα που δεν καλύπτεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. Σχόλια εκτός μικροφώνου. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. Ο κύριος Πρέντα. Επιτρέψτε μου να σας πω κύριε Πρόεδρε, πριν από την τελική ψηφοφορία. Έχουμε μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή από την Επιτροπή ΦΑΜ που είναι 9 παράγραφοι και 45 από τη ΛΥΜΠΕ. Η δική μας είναι 35 μονάχα παράγραφοι. Το κείμενο της ΛΥΜΠΕ είναι πιο μεγάλο από το κείμενο μακροσκελές από το κείμενο της κυρίας Λόγμπιλτερ. Απλό μια παρατήρηση πριν από την τελική ψηφοφορία. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε κατακλειστεί από κείμενα άλλων επιτροπών. Κύριε πρέπει δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας και το είπα προηγουμένω, Θα πρέπει εγκαίρως να πληροφορεί το πρόεδρος για όλα αυτά τα θέματα, τι είναι παραδεκτό και τι δεν είναι παραδεκτό. Και φυσικά και για τις αυτόματες εγκρίσεις θα ήθελα και εγώ να μπορώ να κρίνω για τα θέματα αυτά ή τουλάχιστον πρέπει να συμφωνείτε μεταξύ των συντονιστών. Δεν μπορεί κανείς να γίνει, δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το γιατί υπάρχουν αυτοί οι αυτοματισμοί. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνονται αυτόματες εγκρίσεις και με τον τρόπο αυτό μια έκθεση να περνάει από μια διαδικασία που δεν είναι διαδικασία πολιτικής απόφασης. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και στο μέλλον θα πρέπει να είναι σαφές δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια κρίση για τα θέματα αυτά που είναι θέματα κρίση του εισηγητή και πολιτικής απόφασης. Δεν μπορώ να φαντάζομαι ότι γίνεται μια κρίση για το ότι είναι παραδεκτό για κάτι το οποίο έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα ενδεχομένω. Υπάρχει ένας συντονιστής που έκανε μια ε, παρατήρηση και είχε δίκιο κατά την άποψή μου και ζήτησε το λόγο πριν από την τελική ψηφοφορία. Η δημοκρατία επιτάσσει σε αυτές τις περίπτωσεις να υπάρχει δυνατότητα να ακούσουμε και τις απόψεις από άλλες πολιτικές ομάδες. Και έκανα μία παρατήρηση επί της διαδικασίας, γιατί η διαδικασία που έχει ακολουθεί δεν είναι ικανοποιητική με τις τροπολογίες οι οποίες καλύπτονται ή δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μέρ. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι σωστή διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο Νομίζω ότι είναι σωστό στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να μην υπάρχουν τέτοιες ασάφειες και αβεβαιότητες και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λεχθεί εκπεφρασμένα η κυρία Λοχμπίντερ και θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι σίγουρα είναι πολύπλοκη αυτή η διαδικασία που είχαμε να κάνουμε αλλά η Επιτροπή των Προέδρων των Επιτροπών αποφάσισε ούτω οι επιτροπές, ας πούμε, ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ, ήταν μέρος της διαδικασίας. Αυτή ήταν η απόφαση της συνεδροφής των Πρόεδρων, ώστε να γίνει από κοινού η συζήτηση και με τις επιτροπές ΦΑΜ, ΤΡΟΑ και ΛΥΜΠΕ, και οι οποίες έχουν εν μέρη μια συναρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια δικαιολογία για τα προβλήματα που υπήρξαν, αλλά έχουμε συζητήσει και με τους ε, εισηγητές των ε, επιτροπών αυτών. Αλλά θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι μια έκθεση καταρχήν της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με εξωτερικές σχέσεις καταρχήν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το εξετάσει και πάλι το Προεδρείο μας, αλλά ήταν διαφορετική η απόφαση της, Επιτροπής, της ε, των Προεδρών των Επιτροπών. Σε μια τόσο πολύπλοκη περίπτωση όμως θα ήταν λογικό να συζητήσετε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να τον πληροφορήσετε για τα προβλήματα αυτά, ώστε να μπορέσει το Προεδρείο μας πριν από τη ψηφοφορία που έγινε σήμερα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ψηφίσουμε, τα οποία είναι αναφέρεται ότι καλύπτονται. Για μένα δεν είναι παραδεκτό να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο ένα σφάλμα, λέει ο πρόεδρο. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να είναι σαφέ ότι σε τέτοιες ε, πολύπλοκες περιπτώσεις θα πρέπει η εισηγήτρια ή ο εισηγητής να συνενωθεί και με το Προεδρείο της Επιτροπής του. Τελική ψηφοφορία λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά. Wer dagegen? Wer enthält sich? Αποχές. Aber geschlossen. Mit 44 zu 6 zu 1. 44 με 6 ψήφους κατά και μία αποχή γίνεται δεκτή η έκθεση. Einige kurze Abstimmungen. Με μερικές σύντομες τώρα ψηφοφορίες. Η συμφωνία ευρωμεσογειακή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβάνου Άρχεται την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Σαν τα 6 με 3 εγκρίνεται, συγχαρητήρια, σημείο 7, πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης Λιβάνου για την ε, προσχώρηση Βουλγαρίας Ρουμανίας, ψήφι υπέρ, μάλλον άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά, πέρας. 45 2 1. σε αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Mm? Hm? Do about it? Hm? Ah,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 πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Η συγγήτρια δεν μπορεί να είναι παρούσα δυστυχώς, την αντικαθιστάτε εσείς. Είναι όλα εντάξει, όλα, όλα βαίνουν καλώς. Ψηφίσουμε τότε. Wir kommen jetzt zum Kompromissänderungsantrag 1. Τροπολογία 1 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφεται Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά άποχες έλεγχος. Για την 25. Πέρας. 21 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτή μάλλον απορρίπτεται, αλλά αυτό ελέγξουμε. Πέρας. 29 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Σε διαδίση με τον Πρόεδρο. Πέρας. 36 έξι υπέρ. Επτά κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στο σημείο 10. Πότε θα καταθέσει ο συνάδελφος. Wer macht das? Ich, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einen kurzen... Να σας προτείνω να συζητήσουμε πρώτα το σημείο 12, την ε, αντιπροσωπεία στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, πρωτού καταφτάσει ο κύριος Λερουά εδώ, ο οποίος ε, υποτίθεται θα καταφτάσει ανά πάσα στιγμή στο Σαράγεβο. Πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στη Μόστα. Ο συνάδελφος Πρέντα και ο συνάδελφος Πλένκοβιτς μπορούν ίσως να με ενημερώσουν, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στην αποστολή αυτή. Κάναμε συνομιλίες ε, με τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Α, κατέφτασε όμως ο κύριος Λερουά. Άρα θα ακολουθήσουμε την ε, προβλεπόμενη σειρά των θεμάτων.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 Herzlichen äh, Σα ευχαριστώ και χαίρομαι που είναι εδώ ο Γενικό ε, Διευθυντή τη Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να μα ενημερώσει τι έγινε σε σχέση με το Υπουργικό Συμβούλιο τη χθεσινή ημέρα έγινε μια συζήτηση για την ε, περιφερειακή στρατηγική για το Ιράκ σε ό,τι αφορά την ε, συνάντηση της 17ης Μαΐου στην Βιέννη και του Περιφερειακού Trust Fund και της ε, κρίσης της Συρίας. Όλα τα θέματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά τα 37 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα 21 κράτη-μέλη και την Τουρκία που συμμετέχει προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στο Ιράκ, το Λίβανο και την Ιορδανία. Και επίσης συζητήθηκαν τα θέματα της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Λιβύη, την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ναυτικό και την ακτοφυλακή της Λιβύης. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται με το Ισλαμικό κράτος εκεί σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες του Ισλαμικού κράτους που προτιμάζει από ό,τι φαίνεται νέες δράσεις, νέες ενέργειες εκεί. Και μας απασχολεί αυτό το θέμα, ε, όπως τα θέματα Καθολική στρατηγική και εξωτερική πολιτική. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο. <coughs> Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ εκ μέρου τη κυρία Μογκερίνη, τη είπα τη εκπροσώπου, που έφυγε χθε το βράδυ μετά από το Συμβούλιο για το Μεξικό για να ξεκινήσει τι σημαντικέ διαπραγματεύσει ε, για την ανανέωση τη εμπορική συμφωνία με το Μεξικό. Η συνάντηση χθε ε, ξεκίνησε με την Υπουργική Συνάντηση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Έξι μέλη ήταν παρόντα σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Σκοπός ήταν η αναθεώρηση της πρόοδου μετά από τη Σύνοδο της Ρήγα του Μαΐου 2015. Και μετά ε, είδαμε και την αναθεώρηση του ΕΝΠ e και είδαμε και την αναθεώρηση και την υλοποίηση πώς γίνεται και πώς προχωράει η σταθερότητα στην περιοχή. Να υπενθυμίσω σε όλους, έχουμε την Ουκρανία, την Μολδαβία, τη Λευκορωσία, το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Όλοι συμφώνησαν ότι η συνεργασία ε, στους τομείς που συμφωνήθηκαν στη Ρήγα πέρυσι βαίνουν καλώς. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αντοχή αυτών των χωρών εταίρων. Πολλοί υπουργοί επίσης τόνισαν την ανάγκη να εστιαστούμε στα αποτελέσματα, σε απτά ωφέλη για τους πολίτες όπως η απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ουκρανία και τη Γεωργία και οι ανταλλαγέ ε, φοιτητών και μαθητών και διάφορε άλλε επαφέ για να γίνει πιο αποτελεσματική συνεργασία μα. Είπατε εκπρόσωπο πρότεινε αναθεώρηση τη ε, πολυμερού αρχιτεκτονική ε, ε τη ανατολική εταιρική σχέση. Η επόμενη συνέντευξη θα γίνει το 2017 και θα συμφωνηθεί περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασία μας. Παρό ε, ε, πρόσφατη ε, διένεξη στον ε, Αγκόρνο Καραμπάχ τα πράγματα βαίνουν καλώς και υπήρξε συνένεση για την ενίσχυση της συνεργασίας. Μετά ξεκίνησε το Συμβουλίο και εκεί είχαμε τρία ζητήματα, την περιφερειακή στρατηγική για τη Συρία, το Ιράκ και την μάχη κατά του Νταές, την καθολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μετανάστευση. Θα ξεκινήσουμε τη Συρία. Το Ιράκ και το ΝΤΕΣ ε, είναι μια κοινή στρατηγική. Γνωρίζετε ότι έχουμε μια στιβαρή στρατηγική που υιοθετήθηκε το 2015 για να αντιμετωπίσουμε ολικά τη σύραξη αυτή δεδομένων των ταχαίων εξελίξεων, όπως γνωρίζετε, κάθε έξι μήνες εξολογούν οι υπουργοί τις επιπτώσεις της στρατηγικής και προσαρμόζουν ανάλογα τις προτεραιότητες. Η διαδικασία αυτή εγκρίθηκε χθε με την ε, υιοθέτηση συμπερασμάτων ε, βάσει των οποίων θα συνεχιστούν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ανθρωπιστικά θέματα στη Συρία και στην Ιράκ και εγκριθεί και περαιτέρω δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη Συρία, η κυρία Μογκερίνη έχει δραστηριοποιηθεί στις συνομιλίες ε, της Διεθνούς Ομάδας, ε, ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα στη Βιέννη μαζί με τον απεσταλμένο των ΟΕΕ και με την αντιπολίτευση της Συρίας και έκανε έκκληση προς υπουργού να φροντίσουν να ε, επανεκκινηθούν οι συνομιλίε στη Γενέβη για μια ειρηνευτική μετάβαση το 1η Αυγούστου. Τρεις είναι οι στόχοι. Πλήρης εφαρμογή της εκεχηρίας, ε, πλήρης πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τρίτος στόχος υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης. Αυτά είναι οι τρεις διαδικασίες που υποστηρίζει εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κινητοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από την αρχή τη Συριακή κρίση. Πολλοί υπουργοί κάνουν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στη διαδικασία και η στρατηγική διασφαλίζει ότι θα υπάρχει συμπληρωματικότητα υψηλού επίπεδου βάσει των συμφωνημένων προτεραιοτήτων. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη εμπλοκή και όπω ξέρετε η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, είναι συμπρόεδροι, αλλά και εμείς έχουμε παρουσία και θέλουμε να διδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Επίσης, κυρία Μογκερίνη, ε, τόνισε το κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας στο Ιράκ. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πολιτική στήριξη στην Ιρακινή κυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Επίσης, απαιτείται περισσότερη υποστήριξη από εμάς για τη σταθεροποίηση των απελευθερωμένων περιοχών, για το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και άλλες μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά για το Ιράκ. Η κυρία Μογκερίνη συμφώνησε να καταρτήσουμε επιλογές για την υποστήριξη προς το Ιράκ με του επόμενους μήνες. Όσον αφορά την απειλή του Ντάς, ορισμένοι υπουργοί υποστήριξαν την ενισχυμένη, τον ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην συμμαχία που έχει σχηματιστεί. Αυτά συζητήσαμε στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής και έχουν υιοθετηθεί τα συμπεράσματα φυσικά στα οποία έχετε όλοι ε, πρόσβαση. Ε, στο μεσημεριανό τραπέζι συζητήθηκε η καθολική ε, παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόθηκε ως εντολή στις 15, στον Ιούνιο του 2015 από το Συμβούλιο για να υποβληθεί στο επόμενο Συμβούλιο του Ιουνίου 2016. Βρίσκομαστε σε φάση προετοιμασίας, έγιναν πολλές διαβουλεύσεις. Η κυρία Μογκερίνη ήταν παρούσα εκπρόσωπη του Κοινοβουλίου και η κυρία Μογκερίνη ανέφερε χθε ότι σύμφωνα με την εντολή που έλαβε πέρυσι, τον Ιούνιο του 2015 στο Συμβούλιο, θα παρουσιάσει αυτή την καθολική στρατηγική στο Συμβούλιο 28 και 29 Ιανουαρίου του 2016. Ευρία ήταν η συνένεση των κρατών μελών. Ξέρετε, έχουν γίνει ήδη διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη για τα συνολικά ζητήματα και την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μετά το μεσημεριανό συζητήσαμε, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης. Είναι, φυσικά ότι το θέμα της, είναι φυσικό το θέμα της μετανάστευσης απασχολεί όλους τους υπουργού. Ήταν ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις για τις εξωτερικές πτυχές και ειδικότερα για τους ε, για το διάλογο υψηλού επίπεδου με τις χώρες ε, ε, διέλευσης και προέλευσης και για το πώς η δική μας εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία θα συμβάλλει στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην περιοχή του Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής. Εστιαστήκαμε στα θέματα της επανεισδοχής και του επαναπατρισμού, της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για τις αφρικανικές χώρες με επαρκείς οικονομικούς πόρους, και υποστηρίζοντα το διάλογο με τι αφρικανικέ χώρε, ε, ε, συνοδευόμενο με επενδυτικά πακέτα, ώστε να αυξήσουμε την ε, δυνατότητα επιχειρηματολογία Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι και εκεί συμπεράσματα υιοθετήθηκαν. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα χρησιμοποιηθούν στην, επόμενη, στην επερχόμενη ανακοίνωση για τις εξωτερικές πτυχές της, Ευρωπαϊκής, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση που θα υιοθετηθεί από τους Επιτρόπους στις 7 Ιουνίου, μια κοινή ανακοίνωση για τις εξωτερικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση. Στη συνέχεια συζητήσαμε το μέλλον της επιχείρησης ε, Σοφία, CSDP, στη Μεσόγειο, που αφορά την αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών των ελαφρο, ελαφροδιακινητών ε, ανθρώπων. Το Συμβουλίο κατέληξε σε συμφωνία για τα επόμενα βήματα της επιχείρησης αυτής. Υιοθετήθηκαν συμπεράσματα ώστε να επεκταθεί η επιχείρηση μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Ε, ελήφθη ένα αίτημα από τον Λίβιο Πρωθυπουργό μέσω επιστολής για να προσθεθούν κάποια καθήκοντα στην υπάρχουσα εντολή και τώρα ο επιχειρησιακό προγραμματισμό πρόκειται να ξεκινήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά θα επιταχυνθεί ώστε να εκπαιδευτούν οι συνοριοφύλακε τη Λιβύη και η ακτοφυλακή τη Λιβύη και για τη συμμετοχή στο εμπάργκο των ΗΠΑ ε, για τη Λιβύη και η εντολή θα προσαρμοστεί ανάλογα. Και ξέρετε, γίνεται συζήτηση και στην Νέα Υόρκη για την υιοθέτηση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Ε, τέλος, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, αφορούσαν επίσης την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τον Νότιο Σουδάν, όπου οι καταστάσει είναι πολύ διαφορετικέ, όπω ξέρετε αλλά δύσκολε και στι δύο περιπτώσει. και υπάρχει ε, ε, όλα θα εξερθούν από τις επερχόμενες εξελίξεις. Ε, αυτά συνέβησαν χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και ευχαριστώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Λερουά που μας εξήγησε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω να κάνω μερικά σχόλια. Είπατε ότι συζητήσατε την πρόταση της Κομισιόν για τη φιλελευθεροποίηση ε, προξενικών θεωρήσεων για την Ουκρανία και την Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τι δύο αυτέ χώρε, αλλά και για του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή ΛΥΜΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η αρμόδια επισήλης για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο ποια είναι η δυναμική και τα χρονοδιαγράμματα από την πλευρά του Συμβουλίου για να εγκριθούν οι αρμόδιες προτάσεις, δεδομένου ότι η Ουκρανία επί τη βάση της πρώτης Κομισιόν έχει υλοποιήσει το σχέδιο δράση για τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων και η Τουρκία έχει αναφερθεί σημαντικά ο ρόλος της στον, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές διαστάσεις της πολιτικής μετανάστευσης. Ε, δεύτερο σχόλιο, το σχέδιο δράση για την Συρία και η ανάγκη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μέχρι την 1η Αυγούστου για μια πολιτική μετάβαση μετά από μια μεταβατική περίοδο. Πώς ε, εκτιμάτε τις ε, συνομιλίες της Βιέννης και τις προσπάθειες του Δεμιστούρα και κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό το χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι πολύ κοντά μας η 1η Αυγούστου και έχει μεγάλη σημασία για μας να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα σχετικά. Θυμάμαι κάποτε που το Συμβούλιο αυτό και η, εξωτερική, και η Εξωτερικών αποτελούσαν κάτι που προβαλόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και από τέτοιες ε, συναντήσεις αναμένονταν κάποια αποτελέσματα να προβληθούν κάποια θέματα αλλά αυτή τη φορά πρέπει να παραδεχτώ ότι ναι, ήταν πολύ ωραίο το μέρος όπου πήγα κατά την πράσινη εβδομάδα αλλά δεν ε, πήρα καν χαμπάρι ότι συνέβη αυτή η συνάντηση. Και έχω να σας ρωτήσω το εξή ε, για την ανατολική εταιρική σχέση. Υπό ποιες προποθέσει έλαβε χώρα αυτή η... Τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση όσον αφορά τη σχέση μας με τη Ρωσία. Οι υπουργοί που είχαν κληθεί εκεί τι είπαν. Πώς βλέπουν ε, τις μελλοντικές ε, περιφερειακές και διμερείς σχέσεις τους ε, όσον αφορά τη ρωσική στρατηγική. Και μετά να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πώς τους φαίνεται η κλιμάκωση της ε, στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας ε, στα σύνορα με ορισμένε χώρες και όσον αφορά τις δραστηριότητες με τον ΝΑΤΟ και κάποια ρητορική που ακούμε που όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, μας οδηγεί σε επικίνδυνα νερά. Αναφέρομαι στη ρητορική και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Mr. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια έκθεση όπου αναλύει τι επιχειρησιακέ ικανότητε και αποτελεσματικότητα της UNAFOR ε, της επιχειρήσης ε, Σοφία και είπαν εκεί ότι καταστράφηκαν τα σκάφη ορισμένων λαθροδιακινητών και, αλλά ότι η επιχείρηση υπήρξε αναποτελεσματική στην καταπολέμηση των διακινητών και αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα στους θερμότερους καλοκαιρινούς μήνες όπου η ροή ειδικότερα τώρα των μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα φαίνεται να έχει μειωθεί. Επίσης διάβασα ε, σε εκθέσεις ότι 600.000 μετανάστες αναμένουν σε καταβλισμούς, σε φρικτές συνθήκες στη Λιβύη αφού έχουν αποτελέσει το αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, τοπικών στρατιωτικών δυνάμεων ε, μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιστέλει την ε, δραστηριότητα όλων αυτών των λαθροδιοκινητών που όπως φαίνεται συνεργάζονται με στρατιωτικές δυνάμεις και ενδεχομένως και με το ISIS. Μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι η Λιβύη βάσει της νέας ε, κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα σταθεροποιηθεί και ότι το χάος που εμείς δημιουργήσαμε σε αυτή τη χώρα θα αναστραφεί κάπως γιατί η Λιβύη σίγουρα αποτελεί θέμα ανησυχίας για όλους ε, και ειδικότερα για τους Βρετανούς ε, ενώ επίκειται το δημοψήφισμα. Δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ε, μεταναστών που αναμένουν να έρθουν στην Ευρώπη από τη Λιβύη αποτελεί ένα ζήτημα, ένας παράγοντας που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το δημοψήφισμα της Βρετανίας. Κύριε Φώτηκα, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Λέρο, κύριε Λόχμπίλερ, συγγνώμη. Θέλω να επανέλθω στι εξωτερικέ πτυχέ τη μετανάστευση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που τα περιγράψετε, περιγράφετε και γραπτός πώς θα χρησιμοποιηθεί το Emergency Trust για την Αφρική. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, και αυτό δεν περιλαμβάνεται στα πρακτικά των, συμπερασμάτων του Συμβουλίου, λένε ότι ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων θα έπρεπε προγραμματίστε να δαπανηθούν για την προστασία των συνόρων. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο το θέμα αυτό. Είναι κάποιο σχέδιο που υπάρχει ή απλά κάτι που αναφέρθηκε στα μέσα. Αλλά το διαβάσαμε και στο Σπίγκελ και στο κύριο τηλεοπτικό σταθμό που λένε επίσης ότι οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να το κρατήσουν μυστικό το πού θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα. Και όταν μιλάτε για, διάλογο για στρατηγικό διάλογο πολιτικής με, με χώρες όπως το Σουδάν και άλλες, ε, τίθεται το ερώτημα αυτό, διότι φυσικά οι κυβερνήσεις αυτές έχουν ε, ένα φρικτό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς θα τα λάβετε υπόψη όλα αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πρέντα, έχω δύο σημεία στα οποία, τα οποία θεωρώ ενδιαφέροντα και θα ήθελα κάποια ανάλυση. Πρώτα απ' όλα για την Υπουργική Διάσκεψη με τους Υπουργούς ε, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όσον αφορά τη Μολδαβία διότι στο δελτίο τύπου είδα ένα σχόλιο όπου λέγεται ότι συζητήσαμε για, ένα για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μάθω πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μολδαβία οι υπουργοί διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσει τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως φαίνεται η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ε, απελπιστική εκεί με μια κυβέρνηση που είναι υπέρ της Ευρώπης μένα, αλλά ολιγάρχε. Ε, στη συνέχεια, επειδή το είδα εγώ και το υπογραμμίσετε κι εσείς ε, την ανάλυση της υλοποίησης της συμφωνίας με τους Τούρκους, όσον αφορά τους μετανάστες. Ε, η διένεξη αυτή που σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζεται με τον Ερντογάν στην Τουρκία και η αστάθεια που ε, είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής Πρωθυπουργού θα αλλάξει την εφαρμογή αυτής της, έκθεσης, της συμφωνίας ε, γιατί και γύρω διάφοροι άνθρωποι γύρω από τον Ερντογάν λένε, στέλνουν διάφορα όχι διατραφιλικά μηνύματα, μας λένε ε, ε, βγάλτε εσείς το φίδι από την τρύπα. Ακούμε διάφορα έτσι, μηνύματα πολύ περίεργα από τους ανθρώπους που περιβάλλουν τον Ερντογάν. Ja, dank wel, meneer de voorzitter. Eh, meneer Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λερουά, μία ερώτηση. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου είχαμε ακούσει μία έκθεση για τον πόλεμο στη Συρία και για το Ιράκ και είχαμε μία ανάλυση στην οποία αναφερόταν μία κόκκινη γραμμή. Έχουν τα πράγματα εξελιχθεί. Γνωρίζετε την έκθεση του ΟΗΕ που είναι πολύ αναλυτική και αφορά τα χημικά όπλα είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Οι ειδικέ υπηρεσίε και το Συμβούλιο τι κάνουν όσον αφορά αυτό το θέμα, το εξετάζουν και τι είδου προτεραιότητε αποτελούν τελικά το Ιράκ, η Συρία και τα χημικά όπλα, γιατί τα χημικά όπλα μαζικής καταστροφής είναι αυτά που μα αφορούν, μα απασχολούν περισσότερο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, μια αλυσίδα ολεθρίων ενεργειών. Είναι σκάνδαλο ότι στο Ιράκ εδώ και τέσσερα χρόνια το Ισλαμικό κράτος, το ΝΤΑΕΣ, διατηρεί την οργάνωσή του και την επιμελητία του, η οποία βασίζεται στο εμπόριο πετρελαίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν ποιες είναι οι ευρωπαϊκές, οι διεθνείς εταιρείε οι οποίες έχουν υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπόριο πετρελαίου τόσο προς την κατεύθυνση αυτή και επίσης σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στρατιωτικού υλικού στο Ιράκ. Ποιοι υπέστησαν κυρώσεις για τη Συρία. Το γεγονός ότι έχει εγκαταληφθεί ο ελεύθερος Συριακός στρατός σημαίνει ότι η κοσμική αντιπολίτευση δεν υπάρχει πια στην Συρία με κάποια ισχύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μονάχα τους Κούρδους αποσχιστές, το ΙΠΕΖΕ, Έχουμε το, τον Ασάντ, έχουμε τους Γουαχαμπίτες ακεραιόφρονες και την, ε, το Ντάες. Δεν υπάρχει πια ο στρατός, ο ελεύθερος Συριακός στρατός και η αντιπολίτευση έχουν αποδυναμωθεί τελείως. Και κάνουμε τώρα διαπραγματεύσεις όπου άλλοι έχουν τη στρατιωτική δύναμη και άλλοι αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική εταίροι και έχουμε εγκαταλείψει τελείως τους εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις αυτές της, ε, της ε, Γενέβης. Επίσης η Ρωσία έχει παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στην ενίσχυση του, καθεστώτου του καθεστώτος που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση πριν από δύο μήνες. Επίσης, έχουμε αυτή τη στιγμή εγκαταλείψει τους πρόσφυγες σε καταβλισμούς που βρίσκονται σε πολύ άσχημες συνθήκε είτε στο Λίβανο είτε στα σύνορα της Τουρκίας. Είναι πολύ πιο ακριβό και πολυδάπανο αυτό που κάνουμε από το να είχαμε ενισχύσει αυτούς τους καταβλισμούς στο παρελθόν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και η επιχείρηση Σοφία στην Λιβύη αυτή τη στιγμή, επειδή μίλησα με κόσμο που εμπλέκεται αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση αυτή συνεργάζεται με τις μαφίες που αφήνουν τους μετανάστες 10-15 χιλιόμετρα από τις ακτές Λιβύης και παίρνουν τηλέφωνο τους αρμοδίους στη Σοφία για να τους μαζέψουν. Εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε συνεργοί σε αυτήν τη διακίνηση και διευκολύνουμε τους διακινητές. Στη Λιβύη λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα φάντασμα που θεωρείται ότι είναι η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Κανείς όμως δεν υπακούει σε αυτήν την κυβέρνηση, κανείς δεν υποστηρίζει αυτήν την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα Έχουμε τις πολιτοφυλακές του Σιντάν, της Μισράχα, της ε, Τριπολίτιδος. Δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο η, ο στρατός και κάποιες πολιτοφυλακές σε διάφορες περιοχές της Λιβύης που είναι αυτόνομες και πέραν αυτών των ακυροφρόνων πολιτοφυλακών του Ισλαμικού κράτους. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι με ένα φάντασμα που δεν είναι κυβέρνηση, που προσπαθεί να εξαγοράσει πολιτοφυλακές που δεν το υπακούν καθόλου, θα καταλήξουμε σε μια κυβέρνηση σταθερότητος και ενότητος. Δεν σας μιλάω για τις διαφραγματεύσεις που έχουν γίνει, ούτε για τις ε, δομές που έχουν δημιουργηθεί. Είναι ένα πλασματικό είδο κυβέρνηση στη Λιβύη, με το οποίο πιστεύετε εσεί ότι θα δημιουργήσουμε κάποια ενότητα στη Λιβύη. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος, πάλι δίνει το λόγο. Ο κύριος Μακάλιστερ. Ευχαριστώ. Έχω μια μικρή ερώτηση στην οποία δεν αναφερθήκατε. Οι νέες εξελίξεις στο Ιράν όσον αφορά το άνοιγμα Συγγνώμη, ε, όσον αφορά το άνοιγμα των κεφαλαίων για ε, τη Σερβία, ε, για την προσχώρηση της Σερβίας συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών. Ε, ευχαριστώ και εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα της Λιβύης που έθιξε ο συνάδελφος ο κ. Νάτ. Είπατε ότι έχετε πάρει <clears throat> την εντολή να δημιουργηθεί ε, ένα σώμα ακτοφυλακής, ένα αξιόπιστο σώμα ακτοφυλακής στην ε, Λιβύη. Τι θα κάνουν, θα αναχαιτήσουν τους πρόσφυγες, θα τους στείλουν πίσω στη Λιβύη. Για τι τάξη μεγέθους μιλάμε, για πόσους ανθρώπους, πόσους ανθρώπους έχουμε στη Λιβύη που περιμένουν ή προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι ικανότητες ενός τέτοιου σώματος, ο αριθμός των ανδρών που χρειάζεται για να αναχαιτήσει αυτό το προσφυγικό ρεύμα στη Λιβύη. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι η χώρα αυτή κυβερνάται σε μεγάλο βαθμό από την Αλκάιντα και το ΝΤΑΕΣ και όχι βέβαια από την λεγόμενη <clears throat> κυβέρνηση ενότητος. Πώς μπορείτε λοιπόν να έχετε τη δυνατότητα πραγματικά αυτή η κυβέρνηση να οργανώσει αυτό το σώμα και να αντιμετωπίσει και τις ε, διάφορες αυτές οργανώσεις ε, της ακερόφρονης εκεί. Και η Χωρίς όπλα δεν μπορεί ούτε αυτέ τις, αυτές οργανώσεις να αντιμετωπίσει, ούτε την επιχείρηση σοφία να φέρει σε πέρας. Ποιο είναι ο σχεδιασμό σα, λοιπόν. Δεύτερον, το θέμα των προξενικών θεωρήσεων. Μιλήσαμε για το Κωσυφοπαίδιο, τη Γεωργία, την Ουκρανία και την Τουρκία. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι οι χώρες αυτές έχουν κριθεί βάσει της, των επιτευμάτων τους, βάσει της εκπλήρωσης των προαπαιτουμένων. Θα ήθελα να ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος για την χορήγηση αυτής της φιλελευθεροποίησης προξενικής θεώρησης, ιδίως για τη Γεωργία και το Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τα συμπεράσματα για την περιφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία και το Ιράκ. Το έγγραφο παραθέτει τις προτεραιότητες ε, όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης, ε, σταθερότητας και ασφάλειας. Περιγράφοντας ταυτόχρονα το δράμα ε, των πληθυσμών ε, στις χώρες αυτές και όσον αφορά τις φρεκαλαιότητες που διαπράττει το Ισλαμικό κράτος. Είχαμε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου από το Κοινοβούλιο και που αναγνωρίζει τις φρικαλαιότητες αυτές ως γενοκτονία. Και το ερώτημα μου είναι γιατί οι Υπουργοί Εξωτερικών δεν χρησιμοποιούν την έκφραση αυτή ώστε να αναγνωρίσουν το γενοκτονία. Αν μπορώ να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα, λέω ο πρόεδρος Μπλοκ μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Γκάλερ. <clears throat> Για την Τουρκία παραδείγματο χάρη είναι σαφές ότι η ε, η συγκράτηση του προσφυγικού ρεύματος στις ακτές είναι δυνατή. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό ήδη στις ακτές να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές. Και το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει για τη Λιβύη. Θα ήθελα και εγώ να θέσω το ερώτημα αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ε, η δυνατότητα να πράξουμε κάτι άλλο, πρέπει να έχουμε μία ε, ενέργεια διάσωσης για ανθρωπιστικούς λόγους στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν κάποιοι πρόσφυγες, κάποιοι από αυτούς θα μπορέσουν να περάσουν τους, ε, τα, τον αποκλεισμό αυτό, το οποίο σημαίνει θα πρέπει να θα φτάσουν στην ε, Ιταλία και την Ελλάδα ως πρόσφυγες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια ευρωπαϊκή λύση για το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι πραγματικά πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δύναμη φύλαξη των συνόρων στην Λιβύη κάτω από τις τωρινές ε, ε, συνθήκε η οποία θα είναι σε θέση πραγματικά να δράσει. Ξέρουμε ότι στη σύνθηκε σε άλλα μέρη το Ισλαμικό κράτος είναι ενεργοποιημένο για την διακίνηση ανθρώπων και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια απάντησή σας και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο και κατά πόσο έχει αναφερθεί είτε από το Συμβούλιο είτε από την κυρία Μογκερίνη να υπάρξει και συμπερίληψη της ε, Αιγύπτου στην δύναμη αυτή αναχέτησης των προσφύγων. Ετέθη το θέμα του ρόλου της Αιγύπτου και στην περιοχή της Σύρτης, αλλά γνωρίζουμε ότι υπήρξαν 400 νεκροί που συνελέγησαν στη θάλασσα πριν από δύο εβδομάδες. Αυτοί ξεκίνησαν όχι από το από λιμάνι της Λιβύης, αλλά από την Αίγυπτο. Και ξανάρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια πραγματικά αξιοπρεπή λύση για, την, για το προσφυγικό θέμα. Για μένα αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με τις χώρες οι οποίες είναι όμορες των ακτών από τις οποίες φεύγουν οι πρόσφυγες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιες είναι οι προοπτικές για κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη για την Τουρκία, για την Αίγυπτο και επίσης ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην ε, Λιβύη. Ο κύριος Επιτήριος έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ εάν συζητήθηκε στο Συμβούλιο το τι θα γίνει, πώς αντιμετωπίσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσφυγες από τη Λιβύη. Πού θα τους ε, κατευθύνει τους πρόσφυγες αυτούς, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Οι χώρες αυτές είναι υπερφορτωμένες, δεν μπορούν να αντέξουν άλλους πρόσφυγες θα είναι ουτοπία και όχι σωστή αντιμετώπιση της προκλήσεως εάν πούμε ότι επιτρέπουμε σε κόσμο να φύγει από την Λιβύη ως πρόσφυγες και να πάει στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. Πρέπει να επιλεγεί ένα άλλο μέρος για να πάνε οι πρόσφυγες αυτοί. Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή. thank you very much all for your interest and... Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, προσοχή σας και για τις πολλές και σημαντικές ερωτήσεις που μου θέσατε. Να ξεκινήσω με το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε ότι θα έχουμε τέσσερις υποθέσεις. Στην Ουκρανία, τη Γεωργία, το Κοσμοπέδη και την Τουρκία. Στην ε, ημερησία διάταξη του Συμβουλίου δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ημερομηνίε. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει επί τόπου. Έχουμε μόνο μία συμφωνία με την Τουρκία ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα 72 κριτήρια τα οποία γνωρίζετε όλοι σε ό,τι αφορά την 1η Ιουλίου ε, έχει οριστεί ως ημερομηνία στη Συμφωνία. Φυσικά εφόσον πληρούνται και οι 70 σχετικοί όροι. Δεν υπάρχουν λοιπόν προκαθορισμένες ημερομηνίε. Περίπου την ίδια περίοδο θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις ε, τον Ιούλιο. Δεν έχει οριστεί τίποτα άλλο από το Συμβούλιο. Θα έχουμε Συμβούλιο Τζάε τον Ιούνιο και θα δούμε τι θα αποφασιστεί για τις τέσσερις χώρες. Και για την ε, Λίμπερ. Και πάλι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα δούμε τι θα α, συζητήσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Για τη Συρία. Ε, 1η Αυγούστου για τη μετάβαση έχει οριστεί η ημερομηνία. Κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό ή όχι. Στην Βιέννη του κύριου, με τον κύριο Κάρι ως συμπρόεδρο εξ ονόματος της ομάδας έχει λοιπόν την αίσθηση και εμείς έχουμε την αίσθηση ότι θέλουμε η 1η Αυγούστου να τεθεί ως ημερομηνία προθεσμίας, αν θέλετε, για την πολιτική μετάβαση. Ξέρουμε ότι οι συζητήσει στη Γενέβη δεν ε, πηγαίνουν αρκετά μακριά και χθε το πρωί η κυρία Μογκερίνη συζητήθηκε με τον καινούργιο πρόεδρο Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερω, αλλά ω τώρα Ξέρουμε φυσικά ότι δεν υπάρχει συμφωνία με το ICG για την ε, πολιτική αυτή συμφωνία. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν σαφεί ε, στόχοι, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιτευχθούν. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε και να το προκαταβάλουμε. Για την ε, προσοχή που έχει λάβει στα μέσα ενημέρωση. Στο παρελθόν, ε, ναι, έχει συγκεντρώσει την προσοχή των μέσων ενημέρωση στο FSC, αλλά δεν είναι στόχος μας να συγκεντρώσουμε την προσοχή των μέσων ενημέρωση Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Για την ε, ανατολική εταιρική σχέση, ναι, οι σχέσεις με τη Ρωσία αναφέρθηκαν από, τις, από κάποιες από τις έξι χώρες εταίρους. Μία χώρα όπως ε, η Λευκορωσία είναι ενδιαφέρον ότι αναφέρει, παρόλο ότι εξαρτάται οικονομικά από τη Ρωσία, από τις επιδοτήσεις, από το αέριο, Ξέρουμε ότι χώρες όπως η Αρμενία, η Λευκορωσία έχουν ισχυρούς δεσμούς ε, με την Ρωσία, αλλά παράλληλα θέλουν διακαώς να ε, έχουν πιο πολλέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εταιρική σχέση, το διευκρινίσαμε και χθε, δεν στρέφεται κατά κανενό. Δεν στρέφεται κατά τη Ρωσία, αλλά ο σκοπό έχει να ενισχύσει τι σχέσει με τι έξι χώρε. Η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία έχουν υπογράψει ε, συμφωνία εταιρική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιπε, η Λευκορωσία, η Αρμενία, ε, και οι υπόλοιπε χώρε θέλουν να υπογράψουν τέτοιε συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι τρει λοιπόν θέλουν να υπογράψουν συγκεκριμένες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πνεύμα λοιπόν και πάλι δεν ε, ήταν κατά της Ρωσίας σε καμία περίπτωση. Σχεδόν όλε έχουν ε, πολύ καλές ε, και μάλιστα ε, σχέσεις εξάρτησης με τη Ρωσία, αλλά θέλουν να ενισχύσουν το σκέλος των σχέσεων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήθηκαν θέματα και κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία, θέματα που είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος και για τις έξι αυτές χώρες και θέλουν πραγματικά να έχουν ε, δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά τους ικανοποιεί αυτό τόσο όμορφο τύπο των 28 κρατών μελών με τις έξι χώρες εταιρικής σχέσης. Ε, σε σχέση με τον ΝΑΤΟ τώρα. Στην χτεσινή συνάντηση, όταν συζητήσαμε το θέμα της Ανατολικής ε, ε, γειτονία δεν συμφωνήσαμε, συζήτησαμε το θέμα. Έγινε όμως συνάντηση στο ΝΑΤΟ. Τα 22 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τα άλλα μέλη και έγινε μια συγκεκριμένη συζήτηση σε ό,τι αφορά τη σχέση του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό φυσικά είναι να ενισχυθούν οι σχέσει αυτέ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα το συζητήσουν αυτό το και τον Ιούλιο, ενδεχομένω να υπάρξει μια κοινή συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Θα δούμε κατά πόσον θα προκύψει μια κοινή διακήρυξη, αλλά είναι υπό προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Αναφερθήκατε στην πρόσφατη έκθεση της, ε, για την Ουκρανία Επιχείρηση Σόφια. Προκρίσιμη σημασία. Επιχείρηση Σόφια. Να σα δώσω κάποια εθνικά στοιχεία. Θα θυμάστε καταρχά ότι η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο, λίγε ημέρε μετά το θάνατο 1200 ατόμων στη θάλασσα σε ένα μόνο Σαββατοκυριακό. Ξεκίνησε λοιπόν η επιχείρηση αυτή με βασικό και απότερο σκόπο την καταπολέμηση της διακίνησης ε, ανθρώπων στα διεθνή ίδαντα. Ως τώρα λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε υπόψη μας είναι ότι πάνω από 80 διακινητές έχουν συλληφθεί και πάνω από 100-200 έχουν ε, σταματήσει τις τους. Ξέρετε, αυτό είναι βασικός ο στόχος της επιχείρησης ε, Σοφία και προφανώς ε, υπάρχει Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου στι θάλασσε. Πάνω από 14.000 άτομα έχουν διασωθεί. 14.000 άτομα λοιπόν έχουν διασωθεί από τη θάλασσα. 80 είναι διακινητέ που έχουν συλλεχθεί. Και 14.000 άτομα έχουν διασωθεί. Δεν αρκούν ε, φυσικά αυτά. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα, πολύ παραπάνω. Αλλά είναι ένα επιτεύγμα και πόσοι μετανάστες περιμένουν να έρθουν από τη Λιβύη. Εδώ έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Τα άτομα τα οποία έχουν κατάραχωστεί είναι γύρω στα 10.000, όχι παραπάνω. Ξέρουμε όμως ότι τα αριθμητικά στοιχεία, τα πραγματικά, είναι πολύ πιο υψηλά. Μεταξύ 200 και 80.000 ανθρώπων. Οι πιο πολλοί δεν είναι καν μετανάστες, δεν είναι Λιβύη, είναι αλλοδαποί. Ξέρουμε όμως ότι υπό το Καντάφη υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία πήγαιναν στη Λιβύη για να δουλέψουν. Άρα, πολλά από τα άτομα αυτά, πολλοί από αυτούς τους 200.000, ψάχνουν να βρουν ε, ε, θέσεις εργασίας και αλλού, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνονται συζητήσεις με τον IOM και την υπαδιαρμοστία του, του ΟΗΕ και υπάρχει συνεργασία στη Λιβύη με τοπικούς ε, απασχολούμενους και προσπαθούμε να συζητήσουμε με τα άτομα τα οποία ζουν στους καταβλισμούς αυτούς και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε σε ό,τι αφορά αυτούς που θέλουν να ε, επιστρέψουν στην ε, υπόσαχαρη Αφρική, τι μπορούμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα του καταπιστεύματος για την Αφρική για τη μετανάστευση στο Trust Fund. Αυτό θα θυμάστε ότι δημιουργήθηκε στη Βαλέτα για να βοηθηθεί η αντιμετώπιση των βασικών αιτιών α, της μετανάστευσης και αναφέρθηκε ότι, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν κάποια μυστικά. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Όχι, υπάρχει αυτό το Trust Fund, 1,5 ε, δις ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στα 750.000 ε, ε ευρώ τα οποία έχουν ήδη εκχωρηθεί προ συγκεκριμένου στόχου για την Παλέτα, για την Υποσαχάρη Αφρική, για το κέρα τη Αφρική και πάλι. Έχουν λοιπόν εκχωρηθεί αυτά τα χρήματα ήδη. Αναφερθήκατε σε μυστικά έγγραφα. Δεν υπάρχει τίποτε το μυστικό. Είναι όλα ανοιχτά. Και διαπραγματεύσεις με τις χώρες και η χρηματοδότηση μέσω του Trust Fund. Αναφερθήκατε στο σύμφωνο το οποίο ονομάζουμε ΦΙΣ, το οποίο... Το οποίο συζητήθηκε σε ό,τι αφορά τις 60 χώρες προτεραιότητας. Ενδεχομένω θετικά, αρνητικά κίνητρα για να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση. Αυτό το δελτίο δεν αποτελεί ε, δημόσιο έγγραφο και είδαμε ότι στον Νότιο Σουδάν υπήρχαν κάποιες διαρροές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα οριστικά και φυσικά θα δημοσιευθούν οι σχετικές αποφάσεις. Γίνεται προετοιμασία των συζητήσεων με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον Νότιο Σουδάν και τις άλλες χώρες. Είναι σαφές, απόλυτα σαφές, ότι ενώ εκ παραλίλου θέλουμε να συζητήσουμε θέματα επιστροφών ε, στις χώρες αυτές. Γι' αυτό συμφωνήθηκε και στη Συμφωνία του Κοτονού του άρθρο 13, το οποίο προβλέπει σαφή ε, διαταξή επιστροφής των ε, ατόμων αυτών. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν, δεν αφήνουμε κατά μέρος καθόλου τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό του εγγράφου. Η κυρία Μογκερίνη ε, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Σουδάν πρόσφατα και εκ νέου εξέφρασε ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Το γεγονό ότι υπάρχει η ανησυχία αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συζητήσουμε τίποτα με τη χώρα αυτή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν βασικέ ροέ μέσω Λιβύη, αλλά υπάρχουν και ροέ μέσω τη Νιγηρία. Υπάρχει και ένα ρεύμα μέσω του Νοτιού Σουδάν. Άρα θα πρέπει να συνομιλήσουμε και με το Σουδάν, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο πλαίσιο αυτό. Για τη Μολδαβία μου κάνετε την ερώτηση, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, χθε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δεν συζητήθηκε η εσωτερική κατάσταση στη Μολδαβία διότι δεν αποτελούσε θέμα τη συζήτηση, ε, Συζητήθηκε το σύνολο τη εταιρική σχέση ε, και τα κοινά στοιχεία μεταξύ των έξι χωρών. Αλλά φυσικά η Μολδαβία μα ανησύχει. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι ε, δεν ήταν μόνο χθε το ζήτημα. Σε μια παλιότερη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών είχαμε επισημάνει δύο σημεία πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα. Όταν υπογράφηκε η Συμφωνία Σύνδεσης, διάφορα άνθρωποι από την υπερδνηστερία ζητούν το Μολδαβικό Διαβατήριο για να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο εύκολα. Μας φαίνεται μια καλή μορφή ήπιας πολιτικής και από τότε που υπογράφηκε η εμπορική συμφωνία με τη Μολδαβία διάφοροι επιχειρηματίες από την υπερτρινιστερία ζητούν να υποφεληθούν αυτή τη συμφωνία απελευθέρωση των συναλλαγών για να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας φαίνεται ότι αυτή αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη στη σχέση Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι η εσωτερική κατάσταση όπως είπατε είναι πάρα πολύ δύσκολη και παρότι η κυβέρνηση είναι προευρωπαϊκή, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μετά κάνετε την ερώτηση για τη συμφωνία με την Τουρκία και το πώς αυτό σχετίζεται με τις σημερινές εμπλοκές. Ε, είναι σαφές ότι η στάση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ε, αλλά τελικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα το αποφασίσουν, Όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, θέλουμε να εφαρμόσουμε τα κριτήρια που είχαν προβλεφθεί, να μην αλλάξουν τα κριτήρια αυτά, απλά να τα ε, διεκπαιρεώσουμε πιο γρήγορα ώστε να έχουμε μια απόφαση 1η Ιουλίου. Είναι τα γνωστά 12 κριτήρια, η πολιτική σταθερότητα, ε, η συνταγματική αναθεώρηση δεν ε, υπάρχει εκεί, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης της τρομοκρατίας ναι. Είναι και ένα από τα ζητήματα της συζήτησης σήμερα να δούμε κατά πόσο και ο Σερντογάν θα συμφωνήσει να αλλάξει την νομοθεσία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ή όχι. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι ε, των κριτηρίων αυτών. Αλλά το προεδρικό καθεστώς δεν αποτελεί κομμάτι. Είναι σημαντικό θέμα μένα, αλλά δεν αποτελεί κομμάτι των κριτηρίων που θα εξεταστούν για να αποφασιστεί η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Σας επαναλαμβάνω, θα εξεταστεί αυτό το ζήτημα της απελευθέρωσης, το οποίο, για το οποίο μας ασκούν μεγάλη πίεση, όπως γνωρίζετε. Euh, Τώρα για τα ζητήματα της ε, Συρίας και του Ιράκ. I cannot answer the question of uh, been European beings. Δεν μπορώ να αποφασίσω το ζήτημα αυτό περί ευρωπαϊκών κυρώσεων. Δεν έχω τέτοιε απαντήσεις, αλλά κάνατε διάφορε ερωτήσει ε, για κυρώσεις εγώ δεν έχω απάντηση. Αλλά ε, για την παγκόσμια κατάσταση είπατε ότι έχουμε προβλήματα με την κατάσταση με τη Ρωσία. Ξέρουμε ότι η Διεθνής ε, Συμμαχία συνεχίζει ε, τις εργασίες της. Ε, δεν έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και δεν έχουμε ε, στρατιώτες εκεί στη μάχη, αλλά όπως ξέρετε η Συμμαχία ε, στη Μοσούλη, στη Ράκα. Ε, και οι δύο πόλεις αυτές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια του ΆΙΣΙΣ. Και συζητήσαμε με την Παγκοσμία Συμμαχία ότι ναι, υπάρχει κάποια πρόοδος, αργή μεν, αλλά είναι σαφές ότι η Παγκόσμια Συμμαχία δεν έχει στρατεύματα επιτόπου. Ελάχιστα. Αλλά ευρωπαϊκά στρατεύματα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν ούτε αμερικανικά. Ενδεχομένως κάποιοι σύμβουλοι, οπότε χρειάζεται περισσότερο χρόνος. Η Ρωσία κατέστησε σαφέ ε, ότι ότι το Ιράν έχει εκεί, αυτό είναι αναμφίβολο. Ξέρετε, κερδίζει έδαφο ε, η Παγκόσμια Συμμαχία. Είναι σαφέ ότι κερδίζει έδαφο. Μετά κάνετε μια άλλη ερώτηση για το Σοφία, ότι οι διακινητέ που συνεργάζονται με τη μαφία. Ναι, είναι σαφές αυτό. Η κατάσταση των μεταναστών, των προσφύγων στη Λιβύη, αυτοί που τους βάζουν στη σκάφη, είναι τρομακτική η κατάσταση τους, διότι συχνά μιλάμε για συνεργασία μαφίας και λαθροδιακινητών που τους πιέζουν να μπουν στα πλοία και μεταζητούν χρήματα από τις οικογένειες, από τους συγγενείς. Είναι φοβερή η κατάσταση, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη μας κατά των λαθροδιακινητών. Μετά να αναφέρατε την κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης στη Λιβύη, λέγοντας ότι κανείς δεν τους λαμβάνει υπόψη. Εγώ διαφωνώ, διότι όπως είδατε την περασμένη Δευτέρα στη Βιέννη έγινε μια συζήτηση για να συζητηθεί η Λιβύη και με τις σχετικές χώρες και όλες οι χώρες ε, που έχουν κάποια ε, ενδιαφέρον για το θέμα όπως και η Λιβύη Υπήρχε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΗΠΑ, τη Ρωσία ε, και κατέστησε σαφέ στην διακήρυξη ότι αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση εθνικής συνένεσης ως τη μόνιμη νόμιμη κυβέρνηση, μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Είναι σαφές λοιπόν ότι το κοινοβούλιο του το δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί η πλειοψηφία υπέρ της υποστήριξης αυτής της κυβέρνησης Εθνικής Συνένεσης. Αλλά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αυτού προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει ακόμα να καλέσει το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση. Αυτός ο πρόεδρος ε, είναι ένας από τους τρεις ε, Λίβιους ε, που υφίστανται κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε παρεμποδίζει το σύστημα γι' αυτό το λόγο. Κάτι άλλο πιο ανησυχητικό είναι ότι ο στρατηγός Χαφτά που είναι πολύ σημαντικός έχει πει σαφώς ότι δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης. Οπότε έχουμε συζητήσεις, υπάρχουν επαφές με την Αίγυπτο, αλλά προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί κάτι. Οπότε αποφασίσαμε ότι προς το παρόν η κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης ε, ε, δεν έχει όλες τις εξουσίες που θα έπρεπε να έχει, αλλά είναι η ε, μόνη, νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη. δεν συζητήθηκε η Σερβία ούτε τα νέα κεφάλαια για τη Σερβία. Αλλά η διαδικασία προχωρά μια χαρά. Επίση είναι σημαντικό στο θέμα της Σερβίας να βάλουμε υπόψη και το διάλογο που έχουμε σε υψηλό επίπεδο και με το Κωσφοπέδιο και την Πρίστινα. Όλα αυτά συνεχίζονται, οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία θα ανοίξει και άλλο κεφάλαιο σύντομα. Απλά δεν συζητήθηκε χθε. Το ζήτημα για τη Λιβύη, για την ακτοφυλακή και πώς θα, το, θα δραστηριοποιηθούμε σε όλο αυτό, πώς θα κινηθούμε. Είναι σαφές ότι θα γίνει σε διεθνή ύδατα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αίτημα. Δεν πρόκειται να μπούμε στα ελληνικά εγχωρία ύδατα. Θα μπαίναμε μόνο υπό δύο προϋποθέσεις. Εάν υπήρχε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας βάσει του κεφαλαίου 7, τότε θα είχαμε το δικαίωμα να μπούμε στα εγχωρία ύδατα. Πράγμα πιθανό. Αλλά αυτό που είναι πιθανό είναι ότι σε κάποια φάση η κυβέρνηση της Λιβύας ε, θα μας καλέσει να μπούμε στα εγχώρια ύδατα. Αλλά προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο ούτε στην επιστολή του Προέδρου. Ε, δεν μας ζητά να μπούμε στα εγχώρια ύδατα, οπότε δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα, δεν, μας, δεν έχουμε κληθεί ακόμα. Οπότε όλη η εκπαίδευση θα γίνει στα διεθνή ύδατα με σκοπό ε, τη συνεργασία με τους ακτοφύλακες ε, ώστε να βοηθήσουμε την ακτοφυλακή στην καταπολέμηση του προβλήματος των λαθροδιακινητών. Ε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η διακίνηση ανθρώπων μεταναστών ε, πραγματοποιείται από λαθροδιακινητές, από μαφιόζους που ουσιαστικά πιέζουν αυτούς τους πρόσφυγες να μπουν σε σκάφη για οικονομικούς ε, λόγους και είναι σαφές ότι οι λιβικές αρχές, ε, η κυβέρνηση Εθνικής Συνένεσης και η ακτοφυλακοί θα πρέπει να εργαστούν εντός των εγχώριων υδατών της ε, Λιβύης και εμείς τους υποστηρίζουμε όσο μπορούμε. για την επιχείρηση Σοφία. Βρισκόμαστε στη φάση 2α. Η 2β θα είναι να μπούμε στα εγχωρέδατα και η 2Γ θα είναι πιο κοντά στα λιμάνια. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Χρειαζόμαστε επίσημο αίτημα από τι ελληνικέ αρχέ που ακόμα δεν έχουμε λάβει. Για την Συρία και το Ιράκ. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία αυτά που κάνει το Ισλαμικό κράτο εκεί και το ερώτημα γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτή την φρασιολογία. Οι υπουργοί βέβαια δεν μπορούν να απαντήσουν εξ ονοματό του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δεν χρησιμοποίησε κανένας από τους υπουργού την ε, λέξη γεροκτονία. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω, αυτό θα το πούνε οι υπουργοί. Πρέπει να σας εξηγήσουμε γιατί. Και το ερώτημα του Πρόεδρου Μπροκ. Ναι, είναι σαφές αυτό το οποίο έγινε στην Τουρκία, το συζητήσαμε διάφορες φορές και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων είπε ο Πρωθυπουργό ε, Τσίπρα πώ μπορώ να προστατεύσω τα σύνορά μου εάν δεν συμπεριληφθεί η Τουρκία σε αυτήν τη συμφωνία. Γιατί λίγα χιλιόμετρα μονάχα χωρίζουν τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη από τι τουρκικέ ακτέ. Δεν μπορεί κανεί λοιπόν να προστατεύσει τα εισακτέ χωρί την παρουσία τη ε, Τουρκία. Με την Τουρκία τώρα έχουμε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό μεταναστών που έρχονται για δύο λόγους. Ο κύριος λόγος είναι γιατί, ε, γιατί συνεργάζονται οι, ακτές, οι αρχές της Τουρκίας μαζί μας και γιατί ξέρουν οι μετανάστες ότι δεν είναι τόσο εύκολος ο δρόμος όπως ήταν στο παρελθόν και γι' αυτό έχει μειωθεί η έλευση προσφύγων. Τώρα όμως έχουμε τη συνεργασία των τουρκικών <clears throat> αρχών και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε την ίδια συνεργασία και από τις Λιβικές ε, αρχές. Ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαχράς μίλησε με τηλέφωνο στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και ζήτησε, ήταν παρόν και στην ομάδα υποστήριξης για την ε, Λιβύη και συνεργαζόμαστε μαζί του για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεργασία κατά της μετανάστευσης. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε τη δημιουργία αυτής της ακτοφυλακής και έχουμε και την ε, επιχείρηση ΚΕΠΑ η οποία προετοιμάζεται. Φυσικά δεν θέλει η Λιβύη να έχει στα θέματα ξένα στο έδαφο τη. Είναι μια καθαρά πολιτική επιχείρηση αυτή, ώστε να εκπαιδεύσει τι αστυνομικέ αρχέ και να βοηθήσει την ενίσχυση τη ποινική δικαιοσύνη στην Λιβύη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα των διακινητών προσφύγων. Και το τελευταίο ερώτημα ήταν που θα πάνε οι πρόσφυγες από τη Λιβύη αν έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έρχονται από τη Μεσόγειο πηγαίνουν στις πιο κοντινές χώρες και αυτό σημαίνει Κατάνια, Λαπεδούσα. Ναι, ξέρουμε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνουν τεράστιοι καταβλισμοί προσφύγων. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό προτού φύγουν από τη Λίβη, από τη Λιβύη οι πρόσφυγες αυτοί και θα πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή της χώρας αυτής για να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και γίνονται οι προσπάθειες με το καταπίστευμα για την Αφρική όπως αναφέρατε για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δηλαδή να αποτρέψουμε το να φύγουν αυτοί οι πρόσφυγες από τη Λιβύη και να έρθουν στην Ευρώπη, γιατί η φυσική οδός για αυτούς είναι φυσικά να πάνε από τη Λιβύη στην Ιταλία και η Ιταλία, όπως και οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη προσφυγική ροή. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί η ροή προσφύγων μέσω της κεντρικής Μεσογείου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά για να βοηθήσουμε τις λιβικές αρχές να συνεργαστούμε μαζί τους και η διεγενήση της ακτοφυλακής είναι μοναχα ένα κομμάτι αυτού του εγχείρηματο. Και το δεύτερο τμήμα στην επιχείρηση Σοφία θα είναι να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα έχει η επιχείρηση αυτή την εντολή για την εφαρμογή της, ε, για την εφαρμογή του εμπάργου των ΗΠΑ έναντι της Λιβύης. Ξέρουμε ότι έχουν περάσει διαθαλάσσεις στοιχεία βαριού εξοπλισμού και έχουν καταλήξει στα χέρια της, ε, του Ισλαμικού κράτους, του ΝΤΑΕΣ και γι' αυτό έχουμε αυτό το σχέδιο για να μπορέσουμε μέσω της επιχείρησης Σοφία να εμποδίσουμε την ε, έλευση όπλων και να εφαρμόσουμε το εμπάργο όπλων προς την Λιβύη. Νομίζω ότι προσπάθησα να απαντήσω όλα τα ερωτήματά σας. Για την Αίγυπτο, λέει ο πρόεδρος, η συνέντευξη επιχείρηση Σοφία με την Αίγυπτο, ναι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Πρέπει να συζητήσουμε και με τις Αιγυπτιακές αρχές. Δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για, σε ό,τι αφορά τη Σοφία, αλλά είμαστε πάντα σε επαφή με τις Αιγυπτιακές αρχές, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι κάποια από τα πλοία δεν έρχονται από τη Λιβύη, αλλά από την ε, Αίγυπτο. Αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κράτος στην Αίγυπτο και έχει το, τα μέσα να αποτρέψει τέτοιες ε, ενέργειες και είμαστε σε επαφή μαζί τους για το αν υπάρχει ανάγκη η επιχείρηση Σοφία να επεκταθεί και στην ε, Αιγύπτο βέβαια εάν ε, έρθουν από την Αίγυπτο στις λιβικές ακτές θα παρεμβεί η Σοφία, αλλά δεν έχουμε σχέδια να, γίνει, να επεκταθεί επιχείρηση και στην Αίγυπτο. Και δεν έχω ακούσει τίποτα από τα κράτη-μέλη για μια τέτοια πρόταση. Δεν έχει συζητηθεί λοιπόν το θέμα αυτό. Αλλά ούτε υπήρξε και κάποιο, κάποια προβολή βέτο για την ε, επέκταση μια τέτοια ενδεχόμενη ενέργεια και στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ, ο ευχαριστώ πάρα πολύ. Äh, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το σημείο 11 της ημέρας της διάταξης και έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντεκέρκοφε, ο οποίος είναι συντονιστής για θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμα αριθμίσετε και τα δικά σας τα θέματα, αγαπητοί συνάδελφοι, και καθίσετε στις θέσεις σας, ε, να ξεκινήσουμε και με τα ίσονο σημασία ε, ζητήματα. Κύριε Νάτ, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε παρακαλώ τις συζητήσεις σας. Και χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα. Την τελευταία φορά ήταν τον Ιούνιο του 2015, πριν από 11 μήνες. Και συζητήσαμε θέματα συνεργασίας με τις γειτονικέ χώρες, βάση των όσων είχαν συζητήσει οι Υπουργοί Δικαιοσύνη ε, το Μάιο του 2015. Συζητήσατε και συζητήσαμε θέματα διαλόγου με το Μαρακό και την Τινησία και τα σχέδια διεξαγωγής ε, συζητήσεων με το Λίβανο και την Τουρκία. Και κοιτώντας τις εξελίξεις με τις χώρες αυτές, είναι πιστεύω σοβαρό να συμπεριληφθεί και η διάσταση καταπολέμησης της τρομοκρατία στη συνεργασία με τι χώρε αυτέ. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε με ποιον τρόπο διατέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι προς την κατεύθυνση αυτή. Και το κατά πόσον ε, υπάρχουν θετικές εξελίσεις σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την ειρήνη. Ε, το Συμβούλιο του 21 Απριλίου αποφάσισε να υπάρχει πιο ενσωματωμένη δομή της ανταλλαγής των πληροφοριών στον τομέα της ε, ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και θα θέλαμε να μας πείτε πώς διεξαγόνται οι σχετικές συζητήσεις και κατά πόσο υπάρχουν σχέδια για τις 9 και 10 Μαΐου για το Υπουργικό Συμβούλιο και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε και δύο λόγια για το σχετικό δικό χάρτη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να πάρετε το λόγο και να δημοσιεύσετε τέτοια στοιχεία, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε με ποιον τρόπο ε, οργανώνεται η συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη Europol, η οποία συντονίζει την καταπολίμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο σκοπός της. Ε, αυτό Όμως είναι πραγματική υποχρέωση σε ό,τι αφορά την ε, ε, συνεργασία μέσω της Europol, γιατί έχουμε τις μυστικές υπηρεσίες πέντε χωρών που ακολουθούν τις ε, παραδοσιακές δομές, αν θέλετε, φιλικών μυστικών υπηρεσιών, διμερών δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση. Αυτό θα χρειαζόμαστε, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή σας. Και μετά από τις επιθέσεις ε, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπήρχε επίγνωση του ποιοι κυκλοφορούσαν στα τρομοκρατικά αυτά κυκλώματα, αλλά ενδεχομένω να μην το είχαν μοιραστεί ω πληροφορία και με του άλλου. Και πάντα λοιπόν επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία ότι οι μυστικέ υπηρεσίε λένε ότι τι πληροφορίε αυτέ τι μοιραζόμαστε με όσου εμπιστευόμαστε και μόνο. Και έτσι λοιπόν έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι, επιθέσεις και σε αστυνομικό τμήμα. Ένα άτομο το οποίο, το άτομο μάλλον το οποίο έκανε τις επιθέσεις, ε, είχε εντοπιστεί και είχε ε, εκδοθεί σήμα γι' αυτό τρεις φορές στο κράτος μου, στο κρατήριο της Βασταφαλίας. Άλλε περιστάσει ήταν σαφέ ότι δεν υπήρχε ε, ε, συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, ε, της Γαλλία. Δεν υπήρχε και η σωστή συνεργασία μέσω της Europol προκειμένου τα άτομα αυτά να εντοπιστούν και έτσι έχουμε και τα παραδείγματα τη ελληπού συνεργασία μεταξύ Βελγίου και Γαλλία και χίλια άλλα δυο παραδείγματα. Πείτε μα λοιπόν τι γίνεται. Φυσικά δεσμεύεστε και από το Συμβούλιο, αλλά ε, είσαστε ασφαλώς και Ευρωπαίος και υπάρχουν, ε, λοιπόν, υπάρχει αυτή η έννοια των ευρωπαϊκών ε, θεσμών που θα έπρεπε να συντονίσουν τις δραστηριότητες αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν πιο σύντομος, να αναπτύξω τα διάφορα ζητήματα τα οποία θίξατε και ελπίζω έτσι, να είναι επικοδομητική η συνάντησή μας. Θα ασχοληθώ συνοπτικά με την απειλή και μετά θα αναφερθώ στην απόκριση που έχει αναπτυχθεί από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και το Κοινοβούλιο του τελευταίου μήνε. Και μετά τηλεγραφικά θα αναφέρω ορισμένε από τι ε, προκλήσει που έχουμε να Όσον αφορά την απειλή, ποτέ δεν υπήρξε τόσο σοβαρή όσο Έχω εγώ τη σταδιοδρομία μου εδώ και 18 χρόνια δεν είχα ποτέ να αντιμετωπίσω μια απειλή τόσο οξία και τόσο πολυδιάστατη από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Al-Qaeda ή τον ΤΑΣ, αλλά που εμπνέονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί στη φυλακή. Είναι δύσκολο να οριστεί ο ρυθμός, αλλά είναι υψηλός. Ε, το δεύτερο ανησυχητικό είναι ο αριθμός των αλλοδαπών μαχητών. Έχει μειωθεί μέσα στις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Πιστεύω χάρη στα μέτρα που έχουν λάβει τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και τα κράτη-μέλη. Έχουμε παρατηρήσει σημαντική μείωση, όχι εξάλληψη, αλλά σημαντική μείωση των ανθρώπων που μεταβαίνουν στη Συρία και στο Ιράκ. Και η τρίτη απειλή φυσικά είναι η Αλκάιδα και τον Τάες το ΝΤΑΕΣ όπως γνωρίζουμε παραμένει εντυπωσιακό ως ε, οργάνωση από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων, δυνατοτήτων επικοινωνίας, ε, αριθμό αλλοδοπών μαχητών, αλλά έχει χάσει δύναμη χάρη στις επιθέσεις του συναθλισμού καταπλέμψης του ISIS, ε, χάρη στον Ιρακίνο στρατό, στους Πεσμεργά και άλλες ειδικέ δυνάμεις. Αυτό μπορεί να έχει τρεις συνέπειες ε, όσον αφορά την απειλή. Πρώτον, πρώτη συνέπεια είναι ότι πιθανότατα επιθυμία για επιθέσεις ε, στην, η επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη θα είναι λιγότερες. Ε, ε, είναι κάτι που προβάλλει ιδιαίτερα το ISIS. Είναι πιθανό δηλαδή να σχεδιάσει τέτοιες επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη. Μια δεύτερη απειλή μια δεύτερη απειλή είναι η επιστροφή αλλοδαπών μαχητών πολύ σημαντική σε μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι αναμέναμε και νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Και το τρίτο κομμάτι της απειλής είναι ότι η ηγεσία περνάει από τη Συρία και το Ιράκ στη Λιβύη. Σημαντικά μέλη της ηγεσία. Αλλά να μην ξεχνάμε και την Αλκάιντα, γιατί σε ορισμένου χώρου ε, την ξεχνάμε. Διότι είναι πιο σιωπηλή η Τζαμπατανούστρα Η Τζαμπατανούσα είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι της Αλκάιδα, είναι περίπου... Έχει την ίδια ιδεολογία, ε, διαφορετικές τακτικές από το ΝΤΑΕΣ, αλλά είναι πολύ επικίνδυνος οργανισμός. Αυτά ήθελα να πω για την απειλή. Όσον αφορά την απόκριση μετά τις επιθέσεις του Παρισιού, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Όργανο να κινητοποιηθούν σε τρεις ε, ε, κατευθύνσεις, ε, την ε, αντίδραση προ και μετά των επιθέσεων και η καταστολή. Θέλω να εστιαστώ λίγο στην καταστολή επειδή σας αφορά στις εργασία. εργασίες. Καρδιά των εργασιών μας είναι η βελτιστοποίηση της πλατφόρμας κοινής χρήσης δεδομένων και μου ζητήθηκε από το Συμβούλιο να, αναφέρομαι, να αναφέρω τακτικά στο Συμβούλιο πώς τα κράτη-μέλη ε, παρέχουν στοιχεία και χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες που έχουμε, την Ευρωπόλ που είναι ο βασικός κόμβος ε, ε διαμοιρασμού πληροφοριών, το σύστημα πληροφοριών Schengen που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το πιο αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής που έχουμε που χρησιμοποιούμε εντός ε, της, ε, του χώρου Schengen και μετά έχουμε τη χρήση του Eurodac του συστήματος πληροφορών για τις θεωρήσεις. Έχουμε τη συνεργασία πριν που διασυνδέει τις ε, βάσεις δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα και άλλες πληροφορίες και τα στοιχεία της Interpol. Ε, αυτή την, από αυτή την πλευρά για το SIS ε, έχει βελτιωθεί η χρήση από τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε όπως λέμε διακριτικά τον κόσμο με βάση του άρθρου 36. Πέρασαμε από 1.000 σε 8.000 μέσα σε ελάχιστου μήνες, το οποίο είναι κάτι εξαιρετικό. Όπως είπα, είναι κρίσιμη σημασία σε αυτό για να μπορούμε να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που ε, κινούνται εντό της, ε, ε, του χώρου ελεύθερη μετακίνηση του Σέγγεν. Η Europol ζητά περιθώρια βελτίωση και εμεί το μελετάμε. Η Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου προετοιμάζει ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά, νομικά και κατά κάποιον τρόπο πολιτισμικά εμπόδια ώστε να διαμεριζόμαστε περισσότερες πληροφορίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω περισσότερα αν θέλετε αργότερα. Αυτό αφορά τις δυνάμεις εφαρμογής του νόμου. Έχουμε μια άλλη πρωτοβουλία μεταξύ των ομάδων ε, ασφαλείας. Η αντιτρομοκρατική ομάδα που δημιουργήθηκε μετά ε, την 11η Σεπτεμβρίου έχει αποφασίσει να ενισχύσει τη συνεργασία της και εργάζεται αυτή τη στιγμή στη Χάγη ώστε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανθρώπων και πληροφορικής για μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών με πιο επικοδομητικό τρόπο. Ε, εκεί η πρόκληση θα είναι αργότερα να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ της πλατφόρμας CTG και της ECDC της Ευρωπόλ ώστε να υπάρχει πλήρης ανταλλαγή παντός είδους δεδομένων ε, πληροφοριών που συλλεγεί η Eurojust για παράδειγμα. Οι συζητήσει ε, είναι πολύ εντατικές για αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα τώρα είναι τα σύνορα, στα οποία θα αναφερθώ στο τέλος, αλλά για να αποφύγουμε αυτή την τοξική σύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και μετανάστευσης πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα σύνορα ώστε να, οι χώρες που βρίσκονται ε, πάνω στα εξωτερικά σύνορα, η Ιταλία και η Ελλάδα να είναι εξοπλισμένε με τα απαραίτητα συστήματα ώστε να συλλέγουν ε, δακτυλικά αποτυπώματα και όλα αυτά με την υποστήριξη της Frontex και της Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ αυτή τη στιγμή προσλαμ... προσλαμβάνει ε αξιωματικούς της αστυνομίας οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στα hot spot ε, για ελέγχους. Οπότε τα πράγματα εκεί δείχνουν κάποια βελτίωση. Να μην αναφέρω τι κάνουμε για τα πυροβολά όπλα και τα εκρηκτικά, αλλά είναι σημαντικά ε, και για την καταπολέμηση της χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας. Έχουν γίνει ε, σημαντικά πράγματα. Έχουμε ένα σημαντικό σχέδιο δράση της Επιτροπής, το οποίο τώρα πρέπει να μεταφραστεί σε διάφορα σχέδια νομοθετικά. Τώρα η ποινική δικαιοσύνη είναι κάτι σημαντικό επίση, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε καταδίκε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε σωστά το φαινόμενο. Και το Κοινοβούλιο εδώ θέλει να θετήσει μια οδηγία που θα αφορά όλε τι μορφέ ε, τη τρομοκρατία και του αλλοδαπού μαχητέ. Πρέπει να συλλέξουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό αποτελεί ζήτημα που συζητούμε με τους Αμερικανούς ε, φίλους μας, διότι το, αυτό που συμβαίνει συχνότερα είναι ότι η μόνη αποδείξη που έχουμε είναι ψηφιακή ότι κάποιος πολέμησε με την Αλκάιδα με την Τζαμπατανούσρα. Είναι λοιπόν ε, αποδεικτικά στοιχεία που αποθηκεύονται στην Καλιφόρνια και χρειαζόμαστε ε, αιτήματα μέσω μιας νομικής διαδικασίας που χρειάζεται ένα χρόνο για να πάρουμε την πληροφορία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προσθεθούν και να διευκολυνθούν. Ένα ζήτημα που ακόμα δεν έχουμε συζητήσει στο νέο πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τι αστυνομικέ υπηρεσίε και τι υπηρεσίε ασφαλεία, είναι το ζήτημα τη κρυπτογράφηση. Έγινε μια ζήτηση μεταξύ του CEO τη Apple και του διευθυντή του FBI, θα το ακούσατε, και από αυτό αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση ε, για τι αστυνομικέ αρχέ και τι αρχέ ασφαλεία να έχουν πρόσβαση σε συζητήσει, μηνύματα ε, είναι το θέμα τη κρυπτογράφηση αυτό. Αυτά είναι τα θέματα καταστολή τώρα για την πρόληψη. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις πτυχές το διαδίκτυο, πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε από το δίκτυο το επιβλαβές ε, περιεχόμενο και ξέρετε ότι η Europol έχει δημιουργήσει μια ε, μονάδα που έχει ποσοστό επιτυχίας άνω του 80%. Έχουμε στείλει εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη για να ε, προωθήσουν ε, τη... μια διαφορετική παρουσίαση της, ε, των πραγμάτων αυτών. Όλα αυτά βάσει και τη συμφωνία μεταξύ του Αβραμόπουλου και των εταιριών IT. Κάτι άλλο σημαντικό για όλες τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο θέλουν να έχουν τη δική μας υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί ο διαλόγο με τις εταιρείε, ε, με τις, παροχέ υπηρεσιών διαδικτύου. Το ζήτημα αφορά και την εκπαίδευση των ε, υπευθύνων ώστε να εντοπίζουν τα πρώιμα σημάδια ριζοσπαστικοποίηση. Διότι όσο πιο νωρί εντοπίσει κανεί κάποιο τέτοιο φαινόμενο, τόσο καλύτερη μπορεί να είναι η απόκριση. Έχουμε το σχετικό δίκτυο κατά τη ριζοσπαστικοποίηση, το οποίο εγώ προωθώ γιατί είναι αποτελεσματικό. Αποτελεί άριστη ιδέα τη Κομισιόν και βλέπω ότι όλο και περισσότερες χώρες με ένα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Μια... Τρίτη πτυχή που πρέπει να κάνουμε κάτι <clears throat> και το τονίζω αυτό συνέχεια είναι να δημιουργήσουμε προγράμματα αποκατάστασης. Αυτό αφορά και την Λιβύη και την Τινησία και το Μαρόκο, σε κάποιο βαθμό την Αλγερία. Όλες αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν ένα μεγάλο βαθμό ε, ριζοσπαστικοποίησης. Στην περίπτωση τη Τινησίας έχουμε όχι εκατοντάδες, έχουμε χιλιάδες πολίτες. Δεν μπορεί κανείς να του φέρει όλους αυτούς στο δικαστήριο. Είναι καλύτερα να του βάλει σε ένα πρόγραμμα αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει όμω ότι πρέπει να έχει αναπτύξει ένα ουσιαστικό πρόγραμμα αποκατάσταση. Ξέρω ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και νομίζω ότι το παράδειγμα αυτό πρέπει να έχει μιμητές. Τέλος, οι λεγόμενες ήπιες ενέργειες. Κάτι το οποίο δεν πρέπει <clears throat> να θεωρηθεί ότι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όμως τις απόψεις αυτές στην παιδεία, στο πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ξέρω ότι η κυρία Μογγερίνη ενδιαφέρεται να αναπτύξει την πολιτιστική διπλωματία και εγώ θα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που ήθελε να κάνει ο, και ο πρόεδρος Ομπάμα, να συνδέσει ένα εκατομμύριο πολίτες των ΗΠΑ με πολίτες των αραβικών χωρών μέσω του ίντερνετ. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό και μέσω και του προγράμματος Εράσμους. Αυτό είναι ένα δεύτερο καλάθι πολιτικής και ένα τρίτο το οποίο είναι πιο σημαντικό για την Επιτροπή σας είναι η εξωτερική μας δράση. Θα θυμόσαστε ότι μετά από την επίθεση στο Παρίσι, τις επιθέσεις στο Παρίσι, το Υπουργείο Εξωτερικών μας ζήτησαν να εστιάσουμε περισσότερο στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε αντιτρομοκρατικές εταιρικέ σχέσεις και ενισχυμένο πολιτικό διάλογο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Για αυτή την εταιρική σχέση λοιπόν, το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία μαζί με την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ένωση Ασφαλείας. Η Κομισιόν τονίζει ότι θέλει να πράξει περισσότερο για να δημιουργήσει αυτή την εταιρική σχέση και αυτό είναι θετικό. Μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουμε ένα ουσιαστικό πακέτο μέτρων με την ε, η Ιορδανία, το Λίβανο και την Τινησία. Προσπαθούμε να <clears throat> επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στην ε, περίπτωση της Τινησίας, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική επιχείρηση. Συμφωνήσαμε με τους Τινήσιους φίλους μας σε μια σειρά από στόχους. Δεν θέλουμε μόνο να δώσουμε χρήματα και εξοπλισμό, αλλά θέλουμε όλα αυτά να είναι τμήματα μιας κοινή προσέγγισης για να βελτιώσουμε τη δική τους ανθεκτικότητα στην τρομοκρατία αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας τους να σχεδιάσει <clears throat> μια πλήρη στρατηγική για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Πολλές φορές έχουν μια καθαρά κατασταλτική αντιμετώπιση κατά της τρομοκρατίας με τις δυνάμεις ασφαλείας. Όχι, εμείς θέλουμε να είναι μια πληρέστερη στρατηγική που εμπλέκει όλες τις πτυχές. Παραδείγματος χάρη με τον Πρωθυπουργό της Νησίας συμφωνήσαμε να έχει ένα σύμβουλο εθνική ασφαλείας. Εμεί θα τον βοηθούσαμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να στείλει έξι εμπειρογνώμονε για να υποστηρίξουν τον Σύμβουλο εθνική Ασφαλείας, ώστε και στα κοινωνικά θέματα, στα θέματα τη ε, παιδεία, τη κοινωνία των πολιτών, να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα. Και όχι μονάχα να ασχολείται με τα θέματα ασφάλεια και συνόρων. Δεύτερη πτυχή είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και αυτό έχει τονίσει και ο Οργανισμός Εθνών ότι κάθε μέλος του ΟΗΕ θα πρέπει να δημιουργήσει μία δράση, ένα σχέδιο δράση για την πρόληψη της βίας ενέργειας. Και αυτό πρέπει να κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών και τις γυναίκες κυρίως. Επίσης να υπάρχει μια σαφής προσέγγιση στον τομέα της δικαιοσύνης να ενισχύσουμε τον δικαστικό τομέα, ο οποίος υπάρχει στην περίπτωση της Θυνησίας, ε, αλλά όλοι αυτοί οι συνάδελφοι χρειάζονται πολύ υποστήριξη και εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματικοί. Για τα σύνορα στην, στην, στην ε, Ισία, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί εργάζονται για να βοηθήσουν την Τινησία να εξασφαλίσει τα σύνορα με τη Λιβύη, <clears throat> αλλά έχουμε πολύ περισσότερα που πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι τμήματα μιας πιο πολιτικής συμφωνίας και προσπαθούμε να δούμε όλα αυτά τα προγράμματα ε, χρηματοδότησης, ε, καταπιστεύματα κτλ, την ε, διαδικασία ανάπτυξης, όλα αυτά μπορούμε να κινητοποιήσουμε, τα κινητοποιήσουμε για να επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο που έχουμε, κάνει, που έχουμε συμφωνήσει με την Τινησία και θέλουμε να το επεκτείνουμε αυτό το εγχείρημα και στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Μα ενδιαφέρει πολύ η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, η ασφάλεια των συνόρων. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας. Δεν ξέρουμε τι έγινε με το αεροπλάνο της Egypt το οποίο κατέπεσε. Αλλά αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει όλες τις χώρες τη Μεσογείου να εξασφαλίσουν τα αεροδρόμια και να αυξήσουν την ασφάλεια της αεροπλοίας. Κάποια παραδείγματα των προγραμμάτων που περιμένουμε τώρα να τα εφαρμόσουμε. Ξεκίνησαμε ένα πρόγραμμα 23 εκατομμυρίων στην Τινησία για την μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, εν μέρη για τα σύνορα, εν μέρη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφάλειας για να υπάρχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εποπτεία και συνεργασία με το Υπουργείο ε, Νεότητος και <clears throat> Παιδείας για την πρόληψη στο Ιράκ Έχουμε συμφωνήσει με τον, με τον ε, Σύμβουλο μάλλον Εθνικής Ασφάλειας ένα πρόγραμμα 3,5 ε, εκατομμυρίων να δημιουργήσει μια αρχιτεκτονική για συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση πληροφοριών. Στην Ιορδανία έχουμε ξεκινήσει το μεγαλύτερο προληπτικό πρόγραμμα, 10 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνουμε περισσότερο με την κοινωνία των, πολιτών. Στην Ζάρκα, ιδίω στο βόρειο τμήμα της Ιορδανίας, όπου υπάρχουν ε, Φυλακή ριζοσπαστικοποίηση και επίσης για να αναπτυχθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την πρόληψη. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών και το Βρετανικό Συμβούλιο αναπτύσσουν προγράμματα στο Μαρόκο, το Λίβανο και την ε, Ισία για να ενισχύσουν την κοινωνία των, των πολιτών. Αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν και θα συνεχίσουμε και την εταιρική μας σχέση με το Μαρόκο την Αλγερία και την Αίγυπτο. Είχαμε συναντήσει, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. <clears throat> δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που σα είπα ο Αλέν Λερούα. Κάποια στιγμή η Λιβύη θα είναι στην κορυφή αυτού του καταλόγου για προγράμματα αυτού του είδου. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα μας ζητήσει να ενισχύσουμε τι ικανότητέ τους και φυσικά είμαστε ενεργοί στα Δυτικά Βαλκάνια, το Σλοβενικό Υπουργείο Εσωτερικών πήρε την πρωτοβουλία να φέρει όλους τους εμπλεκομένους γύρω από ένα τραπέζι και μας ενδιαφέρει το θέμα της ε, προ... πρόληψης. Αυτά λοιπόν. Και επίσης όπως μας ζήτησαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, εμπλοκή μας και τον πολιτικό διάλογο με κέρυες χώρες. Για την Τουρκία στις 8 Ιουνίου θα έχουμε μια ειδική συνάντηση για την αντιτρομοκρατία για να αντιμετωπίσουμε πολλές ε, πτυχές μία από τις οποίες είναι πολύ σημαντικές, όπως είδαμε μετά τα δραματικά γεγονότα του Βελγίου, είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ Τουρκίας και εθνικών αρχών, ώστε αν κάποιος επανέρχεται από την Τουρκία στην Ευρώπη να υπάρχει απαραίτητη επικοινωνία. Επίσης, πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Έχω πάει στα Εμμυράτα και στο Κατάρ πρόσφατα και θα πάμε και σε Αραβία πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με, το, με τον κλασικό κόλπο, να τονίσουμε ότι μοιαζόμαστε πάρα πολύ και πρέπει να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ Σαουδικής ε, Αραβίας και του Ιράν. Αυτό είναι και στον πυρήνα των προσπαθειών μας για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στην περιοχή. Πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι και η στρατηγική ασφάλειας για αυτή την περιοχή, για τη Ρωσία. Ξεκινήσαμε κάποιο διάλογο για τα θέματα αυτά με την ε, Ρωσία και έχουμε μετά και το Ιράν. Η ύπατη εκπρόσωπος αποφάσισε να αναπτύξει επιτετραμένους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα γιατί θα έχουμε τώρα άτομα τα οποία θα είναι αρμόδια για να είναι σε επαφή με τους ομολόγους τους, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες και να αναπτύξουμε σχέδια. Κάτι άλλο το οποίο θέλουμε επίσης είναι να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση στα θέματα δικαιοσύνης με την Europol, το Eurojust, με το δίκτυο κατά της ριζοσπαστικοποίηση. γιατί για πολλά χρόνια εμεί ενδιαφερόμαστε μονάχα για την εσωτερική μα ασφάλεια και εστιάζαμε στα θέματα ασφάλεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμω έχουμε φτάσει ένα επίπεδο οριμότητος στα δίκτυα αυτά και έχουμε αυτά τα εξαιρετικά εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να προωθήσουμε μια πλατφόρμα όπω η Europol στι χώρες, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ποινική δικαιοσύνη στις χώρες αυτές της Μεσογείου και το ΣΥΠΟΛ έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για να εκπαιδεύσει είτε στην Ευρώπη είτε στις χώρες αυτές ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και βλέπω πολύ ενδιαφέρον στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για τα θέματα αυτά. Φυσικά θα πρέπει να το θέσουμε αυτό και σε διάφορα πολυμερή φορά. Δεν θέλω να επιστρέψω σε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά την ITC και το σχετικό συνασπισμό. Χθε ε, τονίστηκε ότι θα πρέπει και περισσότερο στι διάφορε ομάδε εργασία να συμμετάσχουμε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη δημοκρατία, τη εγκληματικότητα, τη δημοκρατία για την σταθεροποίηση, την ειρήνη κτλ. Είμαστε μέλο του GCDTF, από ό,τι ξέρετε. του Παγκόσμιου Φόρουμου κατά της Δρομοκρατίας και μία ομάδα εργασία την επόμενη εβδομάδα στο Τσιμπούτι με όλες τις χώρες του κέρδου της Αφρικής θα ε, θέσει τέτοιες διάφορες ε, ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν διάφορα ε, τέτοια κέντρα και διάφορες τέτοιες επιτροπές που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του φόρουμ αυτού και χρηματοδοτούμε όλες αυτές τις δραστηριότητε και προσπαθούμε να τις προωθήσουμε όσο μπορούμε. Στον ΟΗΕ, ασφαλώ, ο Γενικό Γραμματέα προωθεί ένα σχέδιο εργασία το οποίο υποτίθεται θα εγκριθεί τον Ιούνιο. Το υποστηρίζουμε και προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε και για το Κάιρο, όπου και μετέβει, προσπαθούμε να κρατήσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα. Ένα τελευταίο θέμα, φυσικά, περιλαμβάνει την εταιρική σχέση με την ΣΕΙΠΑ. Εγώ στα 22 χρόνια τα οποία έχω δουλέψει σε θέματα ασφάλειας, δεν έχω δει ποτέ σαν η συνεργασία από ό,τι σήμερα. Και νομίζω ότι το κληροδότημα του Σνόουντεν ε, και από διάφορες πρωτοβουλίες, ε, από τα νομοσχέδια για την ε, δυτική σφαίρα, για την Privacy Shield και πραγματικά έχει αλλάξει πορεία ο πρόεδρος Ομπάμα σε σχέση με τον πρόεδρο Μπούς. Άρα το πλαίσιο είναι πολύ καλό και το πρόγραμμα απελευθέρωσης από τις θεωρήσεις που επιτρέπει πάνω από δύο τρίτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνουν στις ΗΠΑ χωρίς θεωρήσεις απασχολεί εν μέρη τις ΗΠΑ. Βλέπουν και την ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση λοιπόν ενδιαφέρονται και έχουν συμφέρον να συμμετέχουν πιο ενεργά γιατί δεν θέλουν φυσικά τρομοκράτε να μεταβαίνουν στι ΕΠΑ. Υποστηρίζουν λοιπόν την Europol σε μεγάλο βαθμό. Πραγματικά θέλουν το σύνδεση e να είναι αποτελεσματικό και η Europol σύντομα θα αναπτύξει πιο στενούς ε, δεσμούς και με το NCDC, το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης ε, της Τρομοκρατίας στη Βιρτζίνια, αλλά και με το FBI. Κατά καιρούς ασφαλώς Έχουμε και διαφορά απόψεων με τη ΣΥΠΑ. Γίνονται συζητήσει για τα ψηφιακά αποτεκτικά στοιχεία, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Θα ήθελα να σα επιστήσω εδώ την προσοχή και στο σχέδιο νομοθεσία, στο νομοσχέδιο που έκρινε την προηγούμενη εβδομάδα η Γερουσία, αν εγκριθεί, θα προκαλέσει σημαντικέ ε, ανησυχίε το Γιάστα σε ό,τι αφορά τους ε, τρομοκράτες και ξέρουμε ότι θα τεθεί βέτο αν εγκριθεί η νομοθεσία αυτή, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτά και τηλεγραμματικά να σας αναφέρω κάποιες προκλήσεις επί τις οποίες θέλω να δραστηριοποιηθώ πιο έντονα. Τι γίνεται με την, το Ισλαμικό κράτος στη Συρία σε ό,τι αφορά τους αεροδόπους μαχητές από την, την Ισία, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και την ανταλλαγή πληροφοριών και ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι η νομοθεσία που ίδρυσε την Europol και την Eurojust είναι τόσο απαιτητική σε ό,τι αφορά το ε, την ιδιωτική σφαίρα που είναι πραγματικά σχεδόν αδύνατον η Europol να έχει ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες αυτές γιατί δεν ε, έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε φανταστοί και φυσικά θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο πολλά μέσω της Interpol σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την τρομοκρατία. Αυτός ο τοξικός σύνδεσμος που μας επιτάσσει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα στα σύνορα, σε ό,τι αφορά επίσης τα πλαστά έγγραφα. Ξέρουμε ότι πολλά έγγραφα τη χάνουν παραποίηση, κλέβονται κτλ. και εξελίξει σε ό,τι αφορά τον τομέα τη ασφάλεια. Πολύ βασικό ζήτημα και αυτό. Και μία πρόσφατη έρευνα σε ό,τι αφορά τι αιτίε ριζοσπαστικοποίηση δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με την ιδεολογία όσο με τη δημοκρατία, την πρόσβαση σε θέσει εργασία, οικονομικέ συνθήκε κτλ. Όσο καλύτερε λοιπόν συνθήκε διαβίωση και εργασία υπάρχουν, τόσο πιο ασφαλή είναι τα πράγματα και πρόεδρε συγχωρέστε με αν μακρηγορίζα. Εκτός του μικροφώνου ο πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιε ερωτήσει όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών πρώτα απ' όλα. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίε. και ξέρουμε ότι αυτό κάνετε εντό των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά η ποσότητα των πληροφοριών δεν ε, χαρακτηρίζει και την ποιότητά τους. Πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι χρήσιμες από όλες αυτές. Θέλουμε να μάθουμε αν με άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει κάποια συνεργασία ώστε να υπάρχουν κάποια κριτήρια ανάγνωσης ώστε να εντοπίζονται οι σημαντικές πληροφορίες. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την εταιρική σχέση με τις χώρες του Περσικού κόλπου, ειδικότερα ε, χώρες που είναι σημαντικές ε, για θέματα πληροφοριών αλλά και για τα θέματα από Ορισμένες από αυτές τις χώρες ήταν οι πρώτες που ε, υιοθέτησαν προγράμματα καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, η Σαουδική τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρα, το Κουβέιτ. Θέλω να μάθω αν προβλέπετε και κάποιες ανταλλαγές με αυτούς, διότι και αυτοί ε, έχουν κάποια τεχνογνωσία και δυνατότητα να παρέμβουν ε, ε, και στο πλαίσιο της Ισλαμικής θρησκείας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συντονιστά, από πλευρά μου πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και να σας ενθαρρύνω για τη δράση σας ε, σε εποχές τόσο δύσκολες. Ε, παρατηρούμε ότι περιγράψετε εδώ όχι μόνο τις δυσκολίες αλλά και τις κατευθύνσεις ε, που θα ακολουθηθούν Δύο σημεία θα ήθελα να τονίσω. Το πρώτο, το τονίσατε και εσείς ε, στην εισαγωγή σας. Επιθυμείτε να ισχυρή ανάπτυξη της προληπτικής πολιτικής ε, για την καταπολέμηση των διαδικτυακών δικτύων ε, στρατολόγησης νέων στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη, και στις αραβικές χώρες. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι συνεργασία σκοπεύετε να αναπτύξετε έτσι με άλλες σχέσεις ε, πέραν των χώρου της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, οι χώρες της Βορειάς Αμερικής. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες φιλοξενούνται σε αυτές τις χώρες. Επίσης, όπως είπε μόλις η κυρία Λιωμαρή, παρατήρουμε ότι αυτή η ριζοσπαστικοποίηση υπάρχει στις αραβικές χώρες αλλά και στις ευρωπαϊκές. στην ε, πολιτική που εφαρμόζετε εσείς υπάρχουν κάποιο είδους συνεργασίες ε, που έχουν προβλεφθεί με τα πολιτισμικά Ισλαμικά κέντρα ώστε σε τελική ανάλυση στην Ευρώπη να ανασχεδιάσουμε την κοινή μας διαβίωση επανεκκινώντας ένα νέο διαθρησκευτικό διάλογο ή προβλέπετε κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες επίσης με οργανισμούς όπως η ΣΕΣΚΟ, Αλέξο, η Ισλαμική Οργάνωση για την Εκπαίδευση της Επιστήμης και τον Πολιτισμό ή τον Αραβικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση και τις Επιστήμες. Ε, οργανισμοί οι οποίοι έχουν κοινά συμφέροντα. με τα ευρωπαϊκά πολιτισμικά κέντρα όπως αυτά που έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες ε, του Μαγκρέπ, του Μασέκ ε, ή στις χώρες του Περσικού κόλπου, όπως μόλις ανέφερε η κυρία Υπουργός Λαλίου Μαρή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα, κύριε Τεκερκόφε, την ε, εκτενή παρουσίασή σας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ένα από τα κράτη που έχει ε, μεγάλη εμπειρία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το αναφέρετε, το Βραϊκό κράτος του Ισραήλ. Και μιλάτε για τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην πρόληψη, σε ό,τι αφορά τις γειτονικές χώρες στην Ιορτανία. Και, κύριε Κεντέχοφτε, ξέρετε ότι Υπάρχει έντονη τέτοια πολιτική και οργάνωση κατά της τρομοκρατίας. Άρα, τι γίνεται με τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας. Και τελευταία ερώτηση. Πρόσφατα δημοσιεύσεις ε, του Ισραηλινού τύπου και των εμπρογνωμόνων τόνισαν την ε, ε, επιτακτικότητα της πυρηνικής απειλής μετά τις φρικτές επιθέσεις των Βρυξελών τίθεται το θέμα και της ε, πυρηνικής απειλής και τα θέματα χημικών όπλων, ε, όπλων μαζικής καταστροφής. Ο πόλεμος στη Συρία αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε χημικό πόλεμο. Πρόκειται πραγματικά για ένα φρικαστικό μελλοντικό σενάριο. Πώς το αντιμετωπίζετε σε ό,τι αφορά δηλαδή, την τρομοκρατία, του κινδύνους της τρομοκρατία, σε ό,τι αφορά το μαζικό επίπεδο, το επίπεδο μαζική καταστροφή ε, βιολογικών ε, όπλων, χημικών όπλων, πυρηνικών όπλων και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ο κ. Αουστροβίτσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίασή σα που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μας παρουσίασε και τις μελλοντικέ γραμμές για τις μελλοντικέ μας δράσεις. Θα ήθελα να υπάρχει όχι μόνο συντονισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση και πιο πολύ κοινή δράση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή μόνο συντονισμό, χρειαζόμαστε και μία συντονισμένη δράση, μία κοινή δράση εξ αρχής. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την αξιολόγησή σας, την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη είναι αποδεκτές αυτές οι πρακτικές ξεπλήματος ε, χρήματος από γειτονικέ κυρίως χώρες όπου υπάρχει πασιφανής πολιτική διαφθορά και όπου τα χρήματα αυτά προέρχονται από βρώμικες δραστηριότητε και τα επενδύουν οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θεωρώ ότι καταρακώνει, θεωρώ ότι καταρακώνει την ε, ε, ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διαφθορά, δεν μπορώ να το ονομάσω αλλιώς. Και αυτό δημιουργεί τεράστιε χρηματοοικονομικέ ροέ, οι οποίε μπορούν να κινηθούν προ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πείτε μας λοιπόν την ε, γνώμη σας. Κάτι άλλο. Μιλήσατε για τη Ρωσία και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Όπως ξέρουμε, στην Τσετσενία ο ηγέτης Καντήροφ διατηρούν 30.000 γραφεία καλά προετοιμασμένα για οποιαδήποτε δράση. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ καλά οργανωμένη οργάνωση και ομάδα. Άτομα τα οποία είναι βετεθειμένα να μεταβούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για να δραστηριοποιηθούν τσετσένοι πολεμιστές οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να περάσουν τα σύνορα του Νότιου Καυκάσου, να πάνε στη Συρία, να διακινήσουν όπλα, να συμμετάσχουν σε πολεμικές δράσεις. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τη συνεργασία ως προς τον κλάδο αυτό, γιατί αυτό αποτελεί μια πραγματική τρομοκρατική απειλή για την Ευρώπη αλλά και για τα άλλα τμήματα του κόσμου και ως εκ τούτου θα ήθελα να μας πείτε τι συμβαίνει από τη δική μας πλευρά στον τομέα αυτό. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια ανερχόμενα μάλιστα φαινόμενα και τέτοιες ανερχόμενες απειλές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Ντικερκόφ, για την ε, ενταλλαχή αυτή παρουσίαση των εργασιών κατά της τρομοκρατίας. Κάποια, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω για να μας πείτε την άποψή σας. Μιλήσατε για του αλλοδαπούς μαχητές. Ότι είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, ότι υπάρχει μείωση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί. Και υπάρχουν ε, και περιστατικά συγκεκριμένες εκτέλεση ε, αλλοδαπών μαχητών με drones. Και υπάρχει και περίπτωση δύο Βρετανών επικών που ε, συμμετείχαν στο Ισλαμικό κράτο ο κ. Ριαδικάν και ο Λιχότ Αμίν, οι οποίοι εκτελέστηκαν από ένοπλο ντρόουν. Πώς αξιολογείτε την περίπτωση αυτή, την υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, έχει ξεκινήσει δικαστική αγωγή. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τη χρήση ένοπλων ε, οχήματων στον αγώνα κατά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρδερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τεκερχόφ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγε εβδομάδε θα αποφασίσουμε αν θα μείνουμε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και δυστυχώ ακούγονται πολλά ε, εκφοβιστικά σχόλια ότι μια έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργήσει διάφορε καταστροφέ ε, και τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ε, απαράδεκτα τα σχόλια αυτά, ειδικότερα δεδομένου των απόψεων που ακούγονται ότι δεν θα υπάρξουν θέματα ασφάλεια. Ε, γιατί μάλιστα η ασφάλειά μα θα βελτιωθεί αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίω και έχει ε, εξελιγμένε υπηρεσίε πληροφοριών και ασφαλεία. Ε, Πολλέ χώρε μάλιστα βασίζονται στι δικέ μα τέτοιε υπηρεσίε σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσετε να συνεργάζεστε με τις Βρετανικές Αρχές διμερώς όπως πράτετε και με άλλα ανεξάρτητα κράτη σε όλο τον κόσμο. Έχετε άλλα σχέδια είδες ε, για τη συγκέντρωση των ε, δυνατοτήτων, των ικανοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής. Συγγνώμη, μπορείτε να μην μιλάτε από εκεί. Ευχαριστώ κύριε Καρβέρ. Δίνω το λόγο στον Αντώνιο Παντσέρη. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Μας περιγράψατε και μας δώσετε μια εικόνα της κατάστασης των εργασιών και της εργασίας με τις διαφορές χώρες, αλλά δεν αναφέρετε μια χώρα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, πρόσφατα υπήρξε μια έρευνα των New York Times Πρόκειται μια χώρα που αποτελεί τη μαύρη τρύπα των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης, το Κωσυφοπαίδιο. Ε, εκεί έχουμε κάποιο είδους κέντρο στρατολόγησης του ΆΕΣΙ στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να καταλάβω, εμείς παρακολουθούμε επαρκώς τη χώρα αυτή και με ποιο τρόπο. Η δεύτερη μου ερώτηση. Πριν λίγες μέρες ε, δολοφονήθηκε με ένα ντρόουν ε, ένας αρχηγός του Ταλιμπάν. Ναι. Ε, και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γενικά οι Ταλιμπάν ε, ήταν περισσότερο, είχαν περισσότερο τοπική και όχι διεθνή δραστηριότητα. Υπάρχει κίνδυνος ε, συγχώνευσης με το ΑΕΣΙΣ και στο Αφγανιστάν με όλες τις συνέπειες που αυτό θα μπορούσε να έχει, όχι μόνο για τη χώρα εκείνη αλλά και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντώνιο. Κύριε Νάρτ, παρακαλώ. Ναι, κύριε Κέρκοφ, τρία ερωτήματα. Καταρχήν, για την ε, για τον προσυλλητισμό στον εξτρεμιστικό Ισλαμισμό, όπω είπατε. Μίλησατε ότι γίνεται αυτό σε μετρεσέδε και σε τζαμιά τα οποία αυτοανακηρύσσονται σε τέτοιου θρησκευτικού φορεί, που κατευθύνονται προ άτομα χαμηλής χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και που λειτουργούν έξω από την παραδοσιακή Ισλαμική κοινότητα. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι παράξενοι φίλοι μας η Σαουδική Αραβία και η χρήση της Τάουα για να διαδώσει τον σαλαφισμό και τον ουαχαμπιτισμό σε άλλες χώρες του κόσμου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι φίλος και σύμμαχος η Σαουδική Αραβία, αλλά παίζει ένα ρόλο προπαγάνδας και προσελθισμού που οδηγεί σε άτομα τα οποία ακολουθούν μια πορεία που είναι, δηλαδή αυτό που τους διαδίδει ακολουθεί μια πορεία τελείως διαφορετική από τον διαφθαρμένο κόσμο της εξουσίας της Σαουδική Αραβία. Με τον τρόπο αυτό δίνουν αυτή την ε, παιδεία μέσα εισαγωγικά στα άτομα αυτά, ώστε να στραφούν κατά της κυριαρχής αρχής. Ένα άλλο πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στην Ισπανία, είναι η πακιστανική, στην πακιστανική του κοινότητα είναι ο δεοβαντισμός που και αυτός προωθεί εξτρεμιστικές τάσεις. Γίνεται κάτι συγκεκριμένο συντονισμού για να αντιμετωπίσετε όχι την Ισλαμική θρησκεία βέβαια, αλλά τον εξτρεμισμό που εκπορεύεται από οργανισμούς που είναι εκτός ελέγχου από την επίσημη θρησκεία. Επίσης, δεύτερο ερώτημα. Η τρομοκρατία έχει σαν στόχο να κτυπήσει με στρατηγικό τρόπο την κοινωνία με την τρομοκράτησή της μέσω μιας ε, ε, τρομοκρατικής ενέργειας που έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό θέλει με, ε, τον τρόπο αυτό να δώσει μεγαλύτερη ε, έμφαση σε θέματα τα οποία κανονικά δεν έχουν κάποια σημασία για ένα πληθυσμό. Στην Μαδρίτη έγινε αυτή η τρομοκρατική ενέργεια πριν από 10 χρόνια, αλλά δεν είχε επιτυχία γιατί δεν μπόρεσε να αλλάξει τους θεσμούς ή τη λειτουργία ενός κράτους. Επομένως, εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό λόγω του συμβολισμού του και το οποίο είναι και προσβάσιμο. Είναι δυνατόν λοιπόν να πετύχει κανείς με ένα σφυρί και με λίγα ε, καλάσνικοφ. Μπορεί κανείς να αγοράσει ένα καλάσνικοφ σε κομμάτια το οποίο μπορεί να γίνει ένα όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε να, άμα το συναρμολογήσει. Με τον τρόπο αυτό είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς μια τρομοκρατική ενέργεια. Εδώ μπορώ εγώ να βγω από τη, στην πλατεία τη, του Λουξεμβούργου, να σπάσω με ένα σφυρί τα τζάμια του κοινοβουλίου, της εισόδου του κοινοβουλίου και να μπω με ένα όπλο και να σκοτώσω μερικούς βουλευτές. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι ευρωβουλευτέ δεν στρέφονται κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι ένα θαυμάσιο στόχο, ο οποίο δεν είναι καν προστατευμένο, γιατί έχουμε φτιάξει αυτέ τι ωραίε πόρτε που ελέγχονται από του ε, φύλακε του κτηρίου, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου είναι πολύ εύκολο να φτάσει κανεί άμα περάσει αυτή την πόρτα. Και εγώ δεν σα τα λέω τώρα επειδή είμαι ιστερικό, είμαι απλό Βάσκο. Είναι προβληματικό για μένα να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Μου φαίνεται σκανδαλώδες ότι εμείς έχουμε κλειστά τα μάτια μας έναντι του μεγαλύτερου τρομοκρατικού στόχου που μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση και γιατί έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Τελευταίο θέμα, η Λιβύη. Μπορεί όλες οι χώρες του κόσμου να αναγνωρίσουν ένα καθεστώς φάντασμα το οποίο του οποίου είτε ένα άτομο το οποίο δεν ξέρει τίποτα. Αλλά η ίδια η Λιβύη δεν, ξέρει, δεν ενδέχεται αυτή την κυβέρνηση. Η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαγοράσει την ε, πολιτοφυλακή της Μιζουράτα και άλλες στη δυτική ζώνη της Λιβύης, πάνω στις οποίες δεν έχει καμία πραγματική δυνατότητα δράσης. Δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο του Χάφερ, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός εταίρος και ε, δύναμη στην ανατολική ε, πτυχή, ούτε αναφέρομαι στον πρόεδρο Αλσάλεχ. Έχουμε στο νότο τις ε, πολιτοφυλακές των Τούμπου, στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της Λιβύης που δεν αναγνωρίζουν κανένα άλλο και δεν αναγνωρίζουν φυσικά, κανείς δεν αναγνωρίζει και τις ε, πολιτοφυλακές των Τουαρέγς που είναι φυλετικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν με τον τρόπο αυτό να έχει ένα αποτελεσματικό αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη Λιβύη. Έχουμε μονάχα ένα καθεστώς το οποίο μόνο μπορεί να ε, δωροδοκεί ε, πολιτοφυλακές για να δράσουν υπέρ του, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει κανεί σε ένα μπορντέλο και να αγοράσει πόνες. Μένετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο αγοράζοντα μισθοφόρου μπορεί κανεί να, ή, να εδραιώσει ένα κράτο. Και πώς είναι δυνατόν επίσης το Ισλαμικό κράτος, το οποίο είναι στην Τέρνα και στη Σύρτη και φυσικά και στο Ιράκ και στη Συρία, πώς μπορεί να έχει κρατήσει αυτή τη βιωσιμότητά του μετά για τόσο μεγάλο χρόνο και που βασίζεται κυρίως στην ε, δυνατότητα διαπερατότητας των, ε, των συνόρων προς το Ιρακίνο Κουρδεστάν, προς την Τουρκία, προς τη Συρία. Πώς είναι δυνατόν αυτό το Ισλαμικό κράτος εδώ και τόσα χρόνια να έχει την επιμελητία, όχι ε, στρατιωτική, αλλά την πρόσβαση σε υλικά πολιτικής χρήσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές χρήσεις. Πώς έχουν χιλιάδες αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα τα οποία είναι στη διάθεσή τους και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Το ίδιο γίνεται και στην Σύρτη και στην Τένα. Γιατί δεν έχει κάνει εμπορίσει κάτι τέτοιο. Κλείνω. Κύριε Κέρκοφ, τώρα ω συνήθω έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε να μας δώσετε τα χρήσιμα στοιχεία και τα ωφέλιμα στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν φαντάζομαι και χθε μεταξύ των Υπουργών σε, ως προς το πώς τοποθετήσετε ε, για θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας, ποια είναι η προτεραιότητα σας κτλ. Ευχαριστώ και να απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν τα ερωτήματα προς την κυρία Μαρή να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι δεν είναι ένα θέμα ποιότητας, είναι και θέμα ποιότητας και αναλυτικής ικανότητα. Νομίζω δε ότι θέτει ένα πραγματικό ερώτημα. Ξέρετε ότι μία από τις μεγάλες δυσκολίες τι οποίε έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα νομική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα πληροφοριών, μυστικών υπηρεσιών και αυτό δεν είναι προσωπική μου απόψη. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθώ να συζητήσω τακτικά. Είχα και συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τους υπεύθυνους των μυστικών υπηρεσιών διαφόρων κρατών ε, μελών, μια γαλλική πρωτοβουλία και νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να ενθαρρύνουμε το εκνητικό ε, πλαίσιο να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τις τέτοιες αναλύσεις μυστικών πληροφοριών. Δεν είναι ρόλος μας ε, προφανώς να το αναλάβουμε εμείς αυτό, αλλά είναι ρόλος μας να ενθαρρύνουμε τους σχηματισμούς αυτούς. Και ξέρω ότι υπάρχει στην Γαλλία μια σχετική ακαδημία για τις μυστικές υπηρεσίες. Ε, το σκέφτονται και οι Γερμανοί. Γιατί να μην υπάρξει λοιπόν ένας ευρωπαϊκός ε, συντονισμός. Ε. Μιλήσαμε για θέματα Five Eyes, πέντε ματιών προηγουμένως. Και όντω η μεγάλη πρόκληση είναι το πώ μπορούμε να αναλύσουμε και να θέσουμε προτεραιότητα στι πληροφορίε αυτέ. Άρα, σίγουρα συμφωνώ και ενθαρρύνω πάρα πολύ αυτή την ιδέα ευρωπαϊκών μυστικών πληροφοριών να υπάρξει δηλαδή και αξιοποίηση των σχετικών πόρων από τον ορίζοντα 2020 και διάφορα από τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνονται στα, στις ανάγκες των συντονιστών. Νομίζω ότι αντιληφθήκατε την σημασία ε, των ε, υπηρεσιών αυτών και το θα πρέπει να τυπώνονται οι ανάγκες τα επόμενα 5, 10 ή 20 χρόνια από τα σχετικά Υπουργεία. Θα πρέπει να διαπιστούν λοιπόν αυτές οι ανάγκες και τίθεται το θέμα ασφαλώς της εσωτερικής ασφάλειας, όπου επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις. Νομίζω ότι αυτή η διάσταση, η πιο αναλυτική λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά την απορριζοσπαστικοποίηση και των ε, εμπειριών που είχαμε στον Περσικό κόλπο και όχι μόνο στον Περσικό κόλπο. Πολλά φυσικά θα πρέπει να ενταχθούμε. γιατί κάποιες εμπειρίες είναι άμεσα χρήσιμες. Για παράδειγμα, ε, επισκέφτηκα το κέντρο απορριζοσπαστικοποίηση στο Ριάντ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακέ οι επιτυχίε που σημειώθηκαν. Και νομίζω ότι υπάρχουν και στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία τέτοια κέντρα, τέτοιε εμπειρίε τι οποίε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θα πρέπει να διαμορφώσει το δικό τη μοντέλο ασφαλώ, γιατί θα πρέπει να λεφθούν υπόψη τρεις παράγοντες ε, σε ό,τι αφορά του αντικειμενικούς παράγοντε, ευαλωτότητα, στόχοι κτλ. Ε, θέματα υποκειμενικά και θέματα ιδεολογικά και θέματα που διευκολύνουν τη διαδικασία και όλα φυσικά εξαρτώνται και από το άτομο και από την, ε, το συγκεκριμένο συγκείμενο. Είναι λοιπόν διαφορετικοί παράγοντες σε κάθε χώρα αλλά σίγουρα συμφωνώ μαζί σας με τη γενικότερη ιδέα ότι θα πρέπει να ενταχθούμε από τις ήδη φυσάμενε εμπειρίε. Για το θέμα του διαδικτύου και το κατά πόσον συνεργαζόμαστε με του εταίρου μα στη ΣΥΠΑ. Ναι, εννοείται, ασφαλώ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητάμε μαζί του Υπάρχει διάσταση και δεν μα ε, χωρίζει μόνο ε, ο Ατλαντικό, αλλά και το First Amendment που μας ε, ορίζει την στάση αυτή και πολλά, κράτα, πολλά κρατημέρια δεν θα μπορούσαν να αποδεχτούν τέτοιες ε, Τι Τίθεται λοιπόν το θέμα λοιπόν του διαδικτύου και οι πιο μικρές ε, χώρες προφανώς έχουν συμφέρον να ενώσουν τις δυνάμεις τους όταν μιλάμε για μεγάλες εταιρείες τύπου Google και τέτοιους κολοσσούς. Χρειάζεται τουλάχιστον ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει ένας διάλογος, πώς να το πω, ισότιμος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, ε, ορίζει μια σχετική στρατηγική Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε ορίσει τις ε, ανάγκες και τις προτεραιότητες, τώρα θα πρέπει να τις διευρύνουμε. Καταρχάς, λοιπόν, θα πρέπει να καταρτήσουμε τις πιο μικρές πλατφόρμες, γιατί όντως το Facebook, το YouTube και η Google έχουν εσωτερικές τέτοιες ικανότητες, αλλά οι πιο μικρές πλατφόρμες δεν διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, ε, ισότητα. Ε, και στο διαφορετική κοινωνία των πολιτών. Το Twitter έχει, για παράδειγμα, ε, μια δυνατότητα ε, εκπαιδευτή των πολιτών, των εργαζομένων σε ό,τι αφορά και την προεκλογική εκστρατεία του Πρόεδρου Ομπάμα στην δεύτερη φορά κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πλανεκτήματα. Το δεύτερο θέμα είναι τα πολιτιστικά ζητήματα. Δεν γνωρίζω όλους τους οργανισμούς που αναφέρατε και θα ενδιαφέρον να τους γνωρίσουμε. Αλλά ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξερευνήσουμε με τους εταίρους μας ε, των αραβικών χωρών πώς μπορούμε από κοινού να προωθήσουμε την διαστρέβλωση, αν θέλετε, του Ισλάμ από από το Ισλαμικό κράτο Και θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά, για την ανάπτυξη ενό ευρωπαϊκού Ισλάμ. Αλλά θα διότι οι πολιτικές μας πούμε σε αυτό είναι διαφορετικέ ε, στην Ευρώπη. Η Γαλλία έκανε για παράδειγμα τη συζήτηση με το Μαρόκο και την Αλγερία για την εκπαίδευση των ημάμιδων. Στην Γερμανία αντίστοιχα υπάρχει μια διαφορετική στάση. Η Αυστρία απαγορεύει την εξωτερική χρηματοδότηση τέτοιων θρησκειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπάρχουν όμως οι όροι για την αναπτύξη ενός Ευρωπαϊκού Ισλάμ. Το ερώτημα του κατά πόσον διεξαγάγεται κάτι παραπάνω από διάλογος και συνεργασία, για παράδειγμα με το Ισραήλ. Ναι. Το ερώτημα του κ. Μπέλτερ δηλαδή. Εγώ έχω μεταβεί διάφορες ε, φορές ε, στο Ισραήλ. Θα ξαναπάω σε ένα μήνα. Διεκταγάγεται επίσημο διάλογο και συζητήσεις για πολλά ζητήματα. Όχι μόνο για τις ε, τρομοκρατικές απειλές, αλλά το πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς για την ασφάλεια των αεροδρομίων και με την Ιορδανία, ασφαλώς. Υποστηρίζουμε μία πρωτοβουλία του βασιλιά της Ιορδανίας για να προωθηθούν ε, ε, με του Ισλάμ από όλες τις ε, ομάδες και ο πρίγκιπας Γκάζη ε, υποστηρίζει πολύ τη διαδικασία αυτή για την ε, πρινική απειλή και τρομοκρατία. CBRN, τρομοκρατία χημική δηλαδή, βιολογική, βιοτεχνολογία. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. Και γι' αυτό τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανοίξει διάφορα κέντρα CBRN σε διάφορα τμήματα του κόσμου, στην Μεσανατολή, στην Ευρωπαϊκή. Είναι ακριβά προγράμματα. Αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για μια ενδεχόμενη απειλή τέτοια φύση. Και θα ήθελα να προσθέσω και την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο αυτό. Μέχρι προσφάτω πίστευα ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά κυβερνοτρομοκρατία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και από αυτή την άποψη. Επί του παρόντο ενδεχομένω να μην αποτελεί εξίσου μεγάλη απειλή, αλλά στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, μπορεί να εξελιχθεί σε τέτοια. Και όχι μόνο η πυρηνική απειλή, αλλά και η χρήση πυρηνικού υλικού γενικότερα για το ερώτημα του κυρίου Άστροβίτσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε κάνει μεγάλη δουλειά για να ε, τροποποιήσουμε, να θεωρήσουμε την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο. Έχουμε την προσέγγιση βάση κινδύνου, risk-based approach, σε ό,τι αφορά και τον εφαρμοστικό κανονισμό για να αντεπίσουμε τις χώρες στις οποίες θα πρέπει να είμαστε πιο ε, προσεκτικοί. Είμαστε σε σωστή λοιπόν ε, τροχιά και θέλουμε να κλείσουμε και τα παραθυράκια της προπληρωμένες ε, κάρτες, τα εικονικά νομίσματα και το καθεξής. Για αυτά που είπατε για την Τζεζανία, δε. Δεν είμαι απολύτως ενημερός για αυτά που αναφέρατε αληθεύει ότι πολλοί πολίτες ε, της Τσετσενίας και του Τζαζιστάν ε, μετέβησαν προς τις κατευθύνσεις αυτές. Ε, και αυτό έχει αντιχτυπώ όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στη Κεντρική Ασία. Γιατί πολλοί από τους πολίτες της Κεντρικής της Ασίας, Τατζικιστάν, Κυργιστάν, Ουσμπεκιστάν, πολλοί εξ αυτών των πολιτών λοιπόν έχουν μεταβεί στην Ρωσία προς εξέβρεση θέσεων εργασία αλλά απολύθηκαν όμω λόγω της οικονομική κρίσης που μας την Ρωσία. Και αυτό προφανώς αποτελεί ένα πόλο ανθρώπων που μπορεί να τους ε, ελκύσει η Συρία. Ακριβώς επειδή υπήρχαν και οι πολεμιστές από την Τσετσενία ε, και τον Δαγκιστάν. Υπάρχουν διαφορέ με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την αντίληψη για τα θέματα αυτά, αλλά προ αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε απόλυτα. Τώρα, για το κατά πόσο αποδέχομαι και υποστηρίζω την χρήση drones ανεπάνδρωτων των τέτοιων ατυχημάτων. Έγινε μια συζήτηση νομική και μη νομική παράλληλα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ επίθεσης από jet fighters και drones από τεχνικής άποψης. Γιατί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σεβαστό ε, το δίκαιο των ε, ένοπλων σειράξεων, το διεθνέ δίκαιο που ορίζουν οι συνθήκε τη Γενέβη. Τώρα, κατά πόσο πρόκειται για ντρόν, ανεπάνδρωτο όχημο ή για ένα πύραυλο που προέρχεται από ένα υποβρύχιο, δεν έχει μεγάλη διαφορά, εξ όσων γνωρίζω. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, στην Συρία, βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε μια ένοπλη σύραξη. και υπάρχει σχετική πρόσκληση από την κυβέρνηση του Ιράκ. Για το ερώτημα του κυρίου Κάρπερ τώρα, για το Brexit. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να ξεκινήσω συζήτηση για το Brexit τόσο λίγο πριν το δημοψήφισμα. Ο Βρετανικός λαός είναι αυτός που θα αποφανθεί. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να μοιραστώ την δική μου εμπειρία. Η Βρετανία συγκαταλέγεται στις χώρες που με βοήθησε πιο πολύ από κάθε άλλη τα τελευταία 8 χρόνια στην καταπολέμηση της τρομοκρατία. Ε, εξ όσων καταλαβαίνω, αυτό σημαίνει ότι η Βρετανία πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει ιδιαίτερο στη διεθνή ασφάλεια ε, το κάνουν προφανώ γιατί είμαι και καλό και ευγενικό και με συμπαθούν, αλλά προφανώ γιατί πιστεύουν και στην προσθέτη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε ασφαλώ όλοι η Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί συνδράμει πολύ στην ιστορική ασφάλεια η Βρετανία και επειδή έχει μακρά εμπειρία στην τρομοκρατία, έχει και πολύ αναπτυχθούν και σύγχρονα συστήματα κατά πολέμηση της τρομοκρατίας στη Βρετανία. Εγώ προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι δεν θα ήταν καλύτερο για την ασφάλεια της, Ευρωπαϊκής, της Βρετανίας να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το κοσυφοπαίδιο εργαζόμαστε για θέματα Δυτικών Βαλκανίων και πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ριζοσπαθικοποίηση σε κάποια από τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και γι' αυτό υποστηρίζουμε απόλυτα μια πρωτοβουλία, όπως είπα και προηγουμένως, ε, του Σλοβενικού κράτους για να υπάρξει συντονισμός ε, των ε, πρωτοβουλειών που βρίσκονται υπό εξέλιξη και στην παρούσα φάση έχουμε δύο-τρεις βασικές προτεραιότητες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα όπλα, τα προβολά όπλα, το τράφικινγκ, τη διακίνηση και το άλλο είναι το στόχο κέρδο της πρόληψης, της για την πρόληψη της ε, στράτευσης. Σε ό,τι αφορά την δολοφονία, την εκτέλεση του αρχηγού του πολεμικού του Ταλιμπάν στην προηγούμενη εβδομάδα, να πω ότι θα πρέπει και εδώ να να ενδυναμώσουμε την κυβέρνηση και να προωθήσουμε μια δικασία ειρήνευση με του Ταλιμπάν. όπω είπαμε, η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι οι Ταλιμπάν μπορούν να ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος του Αφγανιστάν και ξέρουμε πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό. για τον Μοχαμπισμό τώρα και την Σαουδική Αραβία και τον εξτρεμισμό. Συνεργαζόμαστε με την ε, Σαουδική Αραβία για πολλά ζητήματα. Ο πρίγκιπας Βερνέη όταν ήταν ε, υπουργός βοήθησε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και των αλλοδαπών μαχητών είναι πάρα πολύ σε επιφυλακή στο εσωτερικό τη χώρα και θα πρέπει πραγματικά να γίνει συζήτηση αυτή. Σε τι βαθμό δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε την επέκταση του βίαιου σαλαφισμού. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν έχει ρόλο να διαραματίσει στο πλαίσιο αυτό και για το λόγο λοιπόν είπα και προηγουμένω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πιο στενή συνεργασία μα με τη Σαουδική Αραβία για τέτοια ζητήματα. Δεν μπορώ να σχολιάσω το πόσο εύκολο είναι να μπει κανεί εδώ στο κτίριο. Εγώ, τι να σα πω, πέρασα από έλεγχο για να μπω στο κτίριο. Και αυτά τα πρότυπα ισχύουν και για το Συμβούλιο. Ξέρω ότι γίνεται με επαγγελματικό τρόπο αυτή η δουλειά και ένα από του προσωπικού μου bodyguards ήρθε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχει, προσλαμβάνεται πολλούς, είναι καλό αυτό για τη Λιβύη τώρα. Θα πρέπει όντω να αναμείνουμε επίσημη πρόσκληση της, Ευρωπαϊκής, της ε, κυβέρνησης της Λιβύης, της κυβέρνησης Εθνικής ε, Ενότητας. Είμαστε στη φάση εκκίνηση, εκκίνησης. Και ξέρω ότι είπατε ε, εκπρόσωπος ε, θέλει να υπάρξει αυτή η συνεργασία γιατί το Ισλαμικό κράτος απειλεί σοβαρή απειλή για όλες τι γειτονικές χάρες, για τους Σουδανούς, τους Τινήσιους, ε, για τους πολίτες του Σαχέλ τη ε, υποσαχάρης περιοχής και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Γιατί η μισή από τους μάχητες της ΝΤΑΕΣ είναι αλλοδαπή. Και δεν θέλουμε να σχηματιστούν νέα hot spots που θα προσελκύουν τους αλλοδαπούς μαχητές. Διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για μικρό αριθμό, αλλά αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί. Γιατί είναι όλο και πιο δύσκολο να μεταβεί κανείς στη Συρία, γιατί οι Τούρκοι είναι πιο αυστηροί πλέον στα σύνορα. θα πρέπει να προλάβουμε από σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών και να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις να λάβουν γρήγορα δράση και φυσικά είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέρχοφ για τις εκτενείς ε, αναλύσεις. Ε, δυστυχώς όλο και πιο ευαίσθητο γίνεται το θέμα αυτό κάθε χρόνο. Διότι την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ είχαμε πολλές τρομοκρατικές ε, επιθέσεις όχι μόνο στην Ευρώπη δυστυχώς αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, σας ευχαριστώ και έτσι κλείνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Uh, I see that several of our colleagues are waiting. Παρατηρώ ότι πολλοί συναδέλφοι αναμένουν να συζητήσουμε τα επόμενα σημεία, την ενημέρωση με την αντιπροσωπεία Αντόξη, τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη και σχετικά με την πρώτη συνάντηση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εθεροποίηση και Σύνδεση ε, Κωσυφοπεδίου και Παυροβουνίου και την αποστολή τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Αραβική Χερσόνησο στο Κουβέτ και στο Ομάν. Ο κύριο Μπροκ, επειδή βρέθηκε στο Σαράγεβο την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε να αναβάλουμε το σημείο αυτό τη ημερησία διάταξη για την απογευματινό κομμάτι τη συνεδρία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λοιπόν, θα συζητήσουμε αργότερα. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα 12 λεπτά που έχουμε για τα άλλα σημεία, εφόσον συμφωνείτε. Να δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Πετσουλά για την ενημέρωση σε σχέση με το κοσυφοπίδιο και την SAPC. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι όσο πιο σύντομο μπορώ. Στις 17 Μαΐου πήγαμε στην Πρίστινα και δημιουργήσαμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή SAPC ε, για τη σταθεροποίηση και τη σύνδεση. Ε, φτιάξαμε το καταστατικό και τα θέματα τα οποία είναι απαραίτητο να εξετάσουμε για να καταλάβουμε την κατάσταση στο παιδί αυτή τη στιγμή. Να επισημανώ επίσης ότι στις συζητήσεις ε, συμμετείχαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία συνήθως μποϊκοτάρουν τα έργα του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου. Ομόφωνα υιοθετήσαμε κοινέ συστάσεις αλλά η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλού τόνους. Είναι πολλωμένες οι συνθήκες σε θέματα πολιτικές, αλλά αυτό που μας ενθαρρύνει είναι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας βρίσκει σύμφωνη την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και σε αυτό θα πρέπει να βασιστεί η περαιτέρω πολιτική δράση από μέρους μας. Ε, στην επαφή με τα διάφορα πολιτικά κόμματα θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να σταματήσει το σημερινό μπλοκάρισμα του Κοινοβουλίου και να αποφευθούν οι εντάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και επιταχύνει τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις ίδιες δηλώσεις ακούσαμε από όλους τους αξιωματικούς με τους οποίους συζητήσαμε. Τον κύριο Τάτσι, τον κύριο Βέσιλη, τον Πρωθυπουργό Μουσταφά και τον ε, Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Στοιάνοφ. Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ε, τις περαιτέρω δράσεις της ε, Πριστίνα υπέρ του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνάντηση της, η συμφωνία SAPC συζητείται και η απελευθέρωση των θεωρήσεων, οπότε πολύ σύντομα αναμένονται αποτελέσματα όσον αφορά ορισμένα εκκρεμή ζητήματα. πολέμηση τη διαφθορά, του οργανωμένου εγκλήματο, μέσω τη οικοδόμηση ενό πιο αποτελεσματικού δικαστικού συστήματο, συνέχιση τη συζήτηση με τη Σερβία, ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών και τη ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα όλου του βουλευτέ που συμμετείχαν στην ε, Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συνέβαλε ενεργά στην επιτυχία της αποστολής, καθώς και τη Γραμματεία για την εξαιρετική του υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ τον Ιω. Δίνω τώρα το λόγο στον Τον Πρακατσόβιτσα, ε, εκπρόσωπο για το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα και εκ μέρους του κ. Πέτσολα, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ήταν πολύ παραγωγική η εποχή αυτή. Υιοθετήσαμε όλα τα συμπεράσματα ομόφωνα και τον κανονισμό και τις συστάσεις. Έχουν δεσμευτεί για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο για αυτούς αποτελεί ένα στοιχείο συνοχής το οποίο τους ε, συγκεντρώνει όλους μαζί σε κάποιο βαθμό. Οπότε αυτό αποτέλεσε για την αντιπολίτευση μια ευκαιρία ώστε για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό να συμμετάσχουν στις εργασίες ε, του Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Να υπογράμμισω πιο συγκεκριμένα δύο ζητήματα, την απελευθέρωση των θεωρήσεων που αναμένεται, αλλά χρειάζεται να εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικότητα Επίσης είχαμε εκεί και τον Επίτροπο Χάν, ο οποίος ε, επισήμανε τις προϋποθέσεις, ε, δηλαδή το να ρυθμιστεί το ζήτημα του σύνορου με το, Μαυροβού, με το Μαυροβούνιο. Αυτοί δεν το βλέπουν έτσι. Δεν θεωρούν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Ένα δεύτερο ζήτημα που θεωρώ είναι σημαντικό είναι αντιμετώπιση του ζητήματος στο βόρειο Κωσυφοπόδιο, την Ένωση των ε, Σερβικών Δήμων. Η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη διότι δεν μπορούν να υιοθετήσουν ένα καθεστώς βάσει του οποίου η Ένωση των Σερβικών Δήμων θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά όπως φαίνεται αυτό αποτελεί μία από τις προποθέσεις για περαιτέρω διαδικασίες ολοκλήρωσης και ένταξης και πιστεύω ότι θα καταφέρουν τελικά να ε, ε, βρουν μια επιτυχή λύση για αυτό το ζήτημα. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ, η συγγητρία για το Ο και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πράγκα. Και θα ήθελα να συνεχίσω και να συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ήταν καλή επίσκεψη και χάρη και ιδιαίτερα που καταφέραμε σε αυτή την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, σε αυτή την πορεία να υπάρξει αυτή η συμμετοχή και όλα τα γεύματα που διοργανώθηκαν πραγματικά ήταν χρήσιμα και θεωρώ ότι αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενδεχομένως να βοήθησε την απόφαση επιστροφής στις κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Να πω ότι έγινε μια συζήτηση και συνάντηση με τις γυναίκες, τις εκπροσώπους των γυναικών σε ό,τι αφορά των ε, κομμάτων και των Ευρωπών. Ήταν πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Να πω ότι από πλευρά αντιπροσωπείας μας, από τους έξι ευρωβουλευτές, τέσσερις ήταν γυναίκες. Πολύ καλό παράδειγμα θέσαμε, θεωρώ, και να πω επίσης σε ό,τι αφορά το θέμα των συνόρων με το Μαυροβούνιο και της ε, διαχωριστικής γραμμής. υπάρχει έλλειψη κατανόηση για το λόγο, για την αιτία ότι τίθεται αυτό ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, ενώ και άλλες χώρες όπως το Κοσμοπέδιο έχουν τέτοιες διανέξεις με άλλες γειτονικέ χώρες. Γιατί λοιπόν τίθεται αυτό ως όρος για την απελευθέρωση της ε, βίζας. Δεν γίνεται κατανόητο αυτό. Και είναι και δύσκολο να σας πω την αλήθεια να το εξηγήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. <clears throat> Ήταν πράγματι πάρα πολύ καλή αυτή η συνάντηση και υπάρχουν καλές προοπτικές για μεταρρυθμίσεις και πρόοδο στο θέμα της φιλελευθεροποίησης προξενικών θεωρήσεων. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα του σημείου 13 η 12η συνάντηση της Επιτροπής με, την, ε, με το Μαυροβούνιο. Ο ράντο Ράντος θα μας προσθέσει τα πεπραγμένα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω... Μου έχουν ζητήσει να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ε, συνάντησής μας, της Επιτροπής για την Συμφωνία Σύνδεσης. Στην ε, Ποντγκότσα συναντηθήκαμε και προηγουμένως είχε λάβει η χώρα μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας για τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές. Υπήρξε συμφωνία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση κανονικά δεν συμμετέχει στο έργο του Κοινοβουλίου. Δέχτηκε αυτή την απόφαση, αλλά δεν υποστηρίζει συμφωνία για την ε, αναδιάρθρωση τώρα της κυβέρνησης. Έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Μπορεί να κάνει η κυβέρνηση στο χρόνο αυτό που απομένει. Τώρα περισσότερο είναι το θέμα τη εφαρμογή τις ε, πράξεις για τις εκλογές. Πάμε χάρη να μην υπάρξει κρατική χρηματοδότηση υπέρ πολιτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτής. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προσχώρησης, προχωρά με την έγκριση νομοθετημάτων και την ενίσχυση των θεσμών, αλλά το πιο σημαντικό αποτέλεσμα για την εφαρμογή των νέων αυτών μεταρρυθμίσεων είναι ο αγώνας κατά της διαφθοράς και η ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν που πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχουν γίνει δεκτές ομόφωνα αυτές οι συστάσεις. Είχαμε μόνο τέσσερις βουλευτές σε αυτή τη συνάντηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην μεικτή αυτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν δίνει μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου για την Συμφωνία Σύνδεσης με το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ. Και τώρα η Αλβανία. Η κυρία Σλάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αντιπρόεδρο ε, τη αντιπροσωπεία και χρειάστηκε να αντικαταστήσω την κυρία Μακόβα την πρόεδρο, διότι δεν μπορούσε ε, να έρθει αυτή τη φορά. Η συνάντηση έγινε σε μια κρίσιμη εποχή για τη διαδικασία ένταξη τη Αλβανία, όπου η Επιτροπή ΑΝΤΟΚ φτάνει στο τέλο τη ε, δικαστική μεταρρυθμισή που αποτελεί προπόθεση κλειδί για το ανοίγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά και προπόθεση για περαιτέρω πρόοδο των άλλων προτεραιοτήτων, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Το κείμενο μετά από 1,5 χρόνο δουλειά ε, με τη συμμετοχή διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών έχει οριμάσει αρκετά ώστε να μπορέσει να υιοθετηθεί. Παρά του εξαιρετικά πολλωμένου πολιτικού περιβάλλοντος και των πολιτικών εντάσεων στην Αλβανία. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η συνάντηση η CPC έγινε με πολιτισμένο και επικοδομητικό τρόπο. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την τεράστια επιτυχία που έχει επιτευχθεί και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρέστησαν, διότι μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες τις τελευταίες τρεις συναντήσεις, επιτέλους υιοθετήθηκε η κοινή ε, σύσταση με ε, συνένεση αυτή τη φορά. Συζητήσαμε τι τρέχουσε σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αλβανία, τον πολιτικό διάλογο, την πρόοδο σε θέματα δικαστική μεταρρύθμιση, την κατάσταση υλοποίηση του νόμου για την ακαιρεότητα των ατόμων που εκλέγονται σε δημοσιαξιώματα Κάτι που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί επαρκώ, την, εκλο... την μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, κάτι επίση πολύ σημαντικό ώστε να πληρούνται οι συνθήκε για δίκαιε και δημοκρατικέ εκλογέ και φυσικά η μετανάστευση και η περιφερειακή συνεργασία η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης. Οι βουλευτές εστιάστηκαν σε τρία βασικά μηνύματα. Πρέπει να γίνει η δικαστική μεταρρύθμιση χωρίς καθυστέρηση. Είναι σημαντικός ο πολιτικός διάλογος και με το Κοινοβούλιο και η υλοποίηση της ε, νομοθεσίας περί ακαιρεότητας ε, ατομών που εκλεγόνται ή προσλαμβάνονται σε δημοσιαξιώματα. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα ε, υλοποίησης. η πολιτικη ηγέτες ευχαριστα το Κοινοβούλιο για την έκθεση του 2015 για την Αλβανία και επίσης υπόθηκε ότι θα συζητηθεί η γενική πολιτική κατάσταση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία. Όσον αφορά τη γενική πολιτική κατάσταση, η εστίαση ήταν ε, στη δικαστική μεταρρυθμίση και στη νομοθεσία για την αποποινικοποίηση. Οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρθηκαν ε, στην ε, μη εφαρμογή νομοθεσίας και στρατηγικών, την έλλειψη υπηρεσιών σχετικών και επίσημων διαβουλεύσεων που πρέπει να γίνουν όπως και διάφορες άλλες διαδικασίες. Όπως είπα, το μεγάλο επιτέγμα του ACPC ήταν η δυνατότητα μιας φυσιολογικής συζήτησης και η οθέτηση της ε, σύσταση σε αποτέλεσμα απαραίτητης θέσης ε, της αντιπροσωπείας μας από την αρχή της επίσκεψης ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολιτευσή πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να συμφωνήσουν επί ενός κοινού εγγράφου ώστε να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα δεδομένων των τριών τελευταίων αποτυχιών όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση ε, του Κοινοβουλίου για την Αλβανία. Οπότε χρησιμοποίησαμε όλους τους δυνατούς διάβλου για να περάσει αυτό το μήνυμα και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές. Οπότε να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους που ήταν παρόντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σλάιν. Η κυρία Τσέκ θέλει να σχολιάσει ένα σύντομο σχόλιο. Ένα μικρό σχόλιο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να με παρουσιάσει στη συνεδρίαση της Μικρής Επιτροπής, αλλά κάτι το οποίο αναφέρθηκε την προηγούμενη φορά ήταν το θέμα του ποταμού Λιώσα, που είναι ένας από τους τελευταίους ποταμούς στην, ε, στα Βαλκάνια που έχει κανείς δυνατότητα να τον διαπλέψει κανείς με ράφτ με βάρκα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το κομμάτι. Και συναντήκαμε και με τον ε, αναπληρωτή πρωθυπουργό και τους ε, ε, υπενθυμίσαμε ότι η Τουρκία έχει πάρει μια παραχώρηση για να δημιουργήσει ένα φράγμα το οποίο θα πλημμυρίσει όλη την περιοχή. Θέλουμε να του τονίσουμε ότι πρωτού γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει μια ε, έκθεση αντικτύπου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ε, εγγυηθεί αν γίνει μονάχα ένα έργο με την συμμετοχή της Τουρκίας. Δεν πρέπει λοιπόν να καταστραφεί ένας ποταμός ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για το περιβάλλον της ε, Αλβανίας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν Ουλρίκε για το θέμα αυτό και χαιρόμαστε και για την έκθεση της κυρίας Σλάιν γιατί έναντι της τελευταίας έκθεσης που έγινε στο παρελθόν δείχνει ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στο 14ο σημείο την ε, αντιπροσωπεία για την Αραβική Χερσόνησο, Κουβέιτ και Ομάν και δίνω το λόγο στην κυρία Άλλη Ομαρή, την πρόεδρο της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα γρηγορήσω διότι έχουμε ε, πολλά βέβαια. Θέλω να πω στην Επιτροπή ότι χθε μετέβαινε μαζί με τον Ζιλ Παρνιό και την Ελίν Σμιθ την περασμένη εβδομάδα στο Κουβέιτ και στο Ομάν. Αυτή η περιοχή συγκεντρώνει τους περισσότερους ε, κινδύνους ασφαλείας και οικονομίας με τις κρίσεις της Ιεμένης, της Συρίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, της Λιβύης, ε, σημαντικό τρομοκρατικό κίνδυνο και έχουμε και τελευταία και την πετρελαϊκή κρίση. Έτσι λοιπόν το Ομάν και το Κουβέιτ στην περιοχή αυτή, μικρέ χώρε διαδροματίζουν ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Οι συνεδριάσεις ε, που έγιναν στο υψηλότερο επίπεδο με τις αρχές των χωρών αυτών ε, έλαβαν χώρα σε πνεύμα ειλικρίνειας, ε, αμοιβαίου σεβασμού και θα έλεγα μάλιστα και φιλίας. Είναι σημαντικός ο διπλωματικός ρόλος των δύο αυτών χωρών. Μπορέσαμε λοιπόν να διαπιστώσουμε και κάποια συνένεση με τους εταίρους μας όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα των διπλωματικών δράσεων που αυτοί μπορούν να εφαρμόσουν στην περιοχή και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε φώτερε οι πλευρές ότι πρέπει να βρούμε διπλωματικές λύσεις στις ε, σειράξεις της περιοχής. Έτσι λοιπόν επί τη ευκαιρία ε, κάναμε έκκληση για μια πιο στενή συνεργασία και σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών αυτών. Κάναμε έκκληση επίση ε, εκφράζοντα την αναγκαιότητα να κάνουμε και ανακοινώσει για την κοινή γνώμη των χωρών μας ώστε να προχωρήσουν ορισμένα θέματα. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν τρει εβδομάδε στις Βρυξέλλες είχαμε μια πρώτη περιφερειακή κοινοβουλευτική ε, συνάντηση ε, με μεγάλη επιτυχία στις Βρυξέλλες. Αυτή η περιφερειακή διάσταση είναι κάτι νέο στις ε, σχέσεις μας. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι αμοιβέ επισκέψει θα παίξουν σημαντικό ρόλο ώστε να εμβαθύνουμε τι σχέσει μεταξύ των δύο αυτών χωρών ε, του Πεσικού κόλπου ειδικότερα, ώστε να υπάρχει καλύτερη αλληλοκατανόηση. Κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω στα μήμια των χωρών αυτών ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Η επίσκεψή μας καλύφθηκε εκτενώς από τα μέσα των χωρών αυτών, οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέλλον και διάφορες πρωτοβουλίες θα ήταν χρήσιμες. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τις χώρες αυτές του Κουβέιτ, πρόκειται για την 8η ίδια κοινοβουλευτική συνάντηση Συζητήσαμε με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου αυτού και με μέλη της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αλλά μας υποδέχθηκε και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Εμμύρης, ο Αντιπρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισλαμικών Υποθέσεων και ο Υπουργός ε, Εσωτερικής Ασφάλειας και Εσωτερικών με τους συνομιλητές μας ε, ε, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας κοινέ σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας. Επίσης ε, συζητήσαμε για την αναγκαιότητα συντονισμού των προσπαθειών των τοπικών παραγόντων και για τη συμπληρωματικότητα των διπλωματικών δράσεων. Επίσης συζητήσαμε για οικονομικά ζητήματα, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις τις πτώσεις στο τιμό του πετρελαίου στις χώρες αυτές, οικονομικές αλλά και κοινωνικέ. κοινωνικές. Και επί τη ευκαιρία συζητήσαμε και για το θέμα των θεωρήσεων Σέγγεν που για όλες αυτές τις χώρες αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικότερα στο πλαίσιο της διαφοροποίησης και της ε, ενίσχυσης των οικονομικών μας σχέσεων. Είναι και θέμα λίγο πολιτικό, διότι τα τα πέτυχαν ε, χαλάρωση των θεωρήσεων Σέγγεν και αυτές οι χώρες δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτές ε, καθυστερούν τόσο πολύ. Για το διεθνή ρόλο του Κουβέιτ, ε, να υπενθυμίσω ότι στο Κουβέιτ συνεχίζονται οι συνομιλίες ε, για την Ιεμένη υπό την αιγίδα του Οιέ με μια επιτυχία διακοπή των συζητήσεων την ημέρα που εμείς φτάσαμε Ωστόσο η χώρα αυτή θέλει να εμπλακεί ενεργά και υπογράμμισαν το ρόλο τους ε, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Συρία. Επίσης συζητήσαμε εκτενώς για την κατάσταση του, στο Ιράκ και στη Συρία και για την ε, Ισραηλο-Παλαιστινιακή ε, διένεξη και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης του Κουβέιτ υπήρξε αδιάλακτος για το ζήτημα αυτό, είπε ότι η λύση αυτού του προβλήματος είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί οι νέοι άνθρωποι στο Μπεσικό κόλπο να μην γοητεύονται από τα, τρομοκρα... επιχειρήματα των τρομοκρατών και μας ανέφερε μια ιδέα το να αποκλειστεί η Κνεσέτ από την Διεθνή Κοινοβουλευτική Ένωση λόγω μη τήρησης των δεσμεύσεων από το Ισραήλ όσον αφορά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Όσον αφορά το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητήσαμε για την περίπτωση Μπιντούν, για την περίπτωση Μπιντούν. Των Βεδοίνων, ε, ε, ε, ατόμων λοιπόν χωρίς υπηκότητα που βρίσκονται εκεί χωρίς να έχουν υπηκότητα ποιοι εκεί βρίσκονται ως εργαζόμενοι και ποιοι ως ε, ανθρώπους που διαπράττουν απάτη ε, ε προσπαθώντας να, να λάβουν την υπηκότητα για να έχουν κάποια ωφέλη. Επίσης μιλήσαμε για τα μέτρα καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού και για την απορριζοσπαστικοποίηση, διότι και αυτοί έχουν ένα κέντρο το οποίο έφερε προηγουμένως. Όσον αφορά το ΟΜΑΝ, και αυτή ήταν η 8η διακοινοβουλευτική συνάντηση. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο της ε, συνέλευσης και με τον ε, πρόεδρο του, της Γερουσίας, του, αντίστοιχου της ε, σώματος με τη δική μας Γερουσία. Συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό για διάφορα διεθνή προβλήματα και με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Φυσικά συζητήσαμε περί οικονομίας και οικονομικής συνεργασίας. Εκφράστηκε αμοιβή ενδιαφέρον για ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΟΜΑΝ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την διαφοροποίηση των οικονομικών σχέσεων διότι το πετρέλαιο στο ΟΜΑΝ αποτελεί ένα μικρό κομμάτι των δευτεριοτήτων του οπότε συζητήσαμε για το πώς θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις αυτές. Όσον αφορά τα γεωπολιτικά θέματα και τη σχέση με το ΟΜΑΝ και εκεί συζητήσαμε για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και το GCC και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και συζητήσαμε επίσης για το διπλωματικό ρόλο, το σημαντικό διπλωματικό ρόλο που προσπαθεί να διδραματίσει το ΟΜΑΝ στην περιοχή, ειδικότερα όσον αφορά την Εμένη και τη Λιβύη με όλες τις δυσκολίες που το υπογραμμίζω που αυτό συνεπάγεται στη σχέση με την ε, Σαουδική Αραβία και το Ομάν είναι η χώρα που μας φαίνεται να ε, είναι πιο κοντά στο Ιράν να έχει ένα πιο, ε, πιο βαθύ διάλογο με το Ιράν το οποίο του δίνει τη δυνατότητα διάλογο με το Ιράν το οποίο φυσικά οδηγεί σε κάποιε επιφυλάξει ε, προ το ΟΜΑΝ από άλλε χώρε όπω η Σαουδική Αραβία. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όχι μονάχα το να επισκεπτόμαστε και να συζητάμε, αλλά να δούμε τι θα γίνει για όλα αυτά τα θέματα. Εμείς θα έχουμε και μία συνάντηση όλων αυτών των χωρών εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 και έχουμε προτείνει να προετοιμαστούμε με διάδες ουσιαστικά κοινοβουλευτικών και πολιτικών υπευθύνων που θα εργαστούν από κοινού μέσω του διαδικτύου για συγκεκριμένα θέματα, ώστε να μπορούμε να έχουμε συζητήσει επί συγκεκριμένων θεμάτων. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το διακοινοβουλευτικό διάλογο σε διμέρε επίπεδο. Εγώ έχω προσκαλέσει τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων του Κουβέιτ και τον ε, Αντιπρόεδρο, τον μάλλον τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Πρωθυπουργό του Ομάν να έρθουν για να μιλήσουν ενώπιον τη Επιτροπής μα, Έχω προτείνει επίση να υπάρξει και μία επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ για να προετοιμάσουμε και τη διαδικασία των συμφωνιών επένδυση Ευρωπαϊκή Ένωση Ομάν και Ευρωπαϊκή Ένωση Κουβέιτ. Είναι μια πολύ σημαντική λοιπόν ε, πρόταση να οργανώσουμε και ένα σεμινάριο για του εκπροσώπους των μέσων ενημέρωση αυτών των χωρών εδώ για τη δική μας εικόνα και για τη συνέχεια των προσπαθειών μας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Ήταν πολύ θετικά αυτά. Χαίρομαι που ήταν χρήσιμε οι επισκέψει στο Κοβέιτ και στο Ομάν για την συνειδητοποίηση κυρίω των πληθυσμών εκεί για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σα. Επίση είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που προτείνεται για τα μέσα ενημέρωση. Τούτων λεχθέντων μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση του πρωινού. Ξεκινάμε και πάλι στις 3 ε, η ώρα. Και θα είναι και ο πρόεδρος Μπρόκ, ίσως.